Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας θα μπορούσαμε να αρχίσουμε παρακαλώ με την έγκριση του σχεδίου ημερησίας διάταξης. Θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή πολιτική για την ε, Διαρθρητική πολιτική και την πολιτική συνοχή. Θα προσθέσουμε ένα νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη μετά το 10, πριν από τα 11, τα διάφορα. Θέμα που έχει σχέση με την παρουσίαση από τους συντάξτες μια σύντομη ομιλία για τα μέσα για την διαχείριση της αλίας. Επίσης ζητήθηκε από την κυρία Ροντόστ να προσπαθήσουμε να βρούμε χρόνο σήμερα για να συζητήσουμε το θέμα της πετρελαιοκυλίδας στον κόλπο του Μεξικού και τις επιπτώσεις που ενδεχομένω θα μπορούσε να έχει στην Αλία. Νομίζω ότι πρόκειται για πολύ καλή υπόδειξη. Ήρθαμε σε επαφή χθε το βράδυ με την Επιτροπή όταν η κυρία Ράντα έκανε το αίτημα αυτό που μας είπε ότι ακόμη δεν είχαν αρκετό χρόνο να στείλουν από την ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος εμπειρογνώμονα. Δεν θέλω να προτείνω ότι αν έχουμε χρόνο στο τέλος της ε, σημερινή ημερησία διάταξη σήμερα το πρωί να έχουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας και να ζητήσω στην ε, επόμενη συνεδρίαση να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό με έναν πραγματογνώμονα από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, από την Επιτροπή για να μας ενημερώσει. Αν δεν έχουμε χρόνο σήμερα το πρωί θα πρότεινα να βρούμε χρόνο σήμερα το απόγευμα αν ε, έχουμε χρόνο προς το τέλος του της Κύριε Ρόντο, λοιπόν, θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων, εάν ε, συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Τώρα, σας πω ότι θα ψηφίσουμε, όπως ξέρετε, σήμερα το πρωί θα τις κάρτες σας, κάτι ψηφοφορίες. Εάν την έχετε ξεχάσει, να προσπαθήσετε να την βρείτε τον συντομότερο δυνατό. Επίσης πρέπει να πω ότι μεταδίδεται απευθεία από το ίντερνετ η συνεδρία. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης. 15 και 16 Μαρτίου, ως συνήθως, εάν μέχρι το τέλος συνεδρίας δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα θεωρήσω ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Ανακοινώσει του Προέδρου. Στο σημείο 3, όπως γνωρίζετε, Δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που αφορούν την μεταρρύθμιση κοινή ελληνική πολιτική οργανώθηκαν αυτή την αυτή εβδομάδα από την Ισπανική Προεδρία στη Γαλλικία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό εξηγείται σήμερα και από δύο συναδέλφων. Η πρώτη συνεδρία αφορά την πολιτική ελεία τη Δευτέρα και τη Μαΐου στην ε, Λακορούνια, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200 συμμετέχοντε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τι εθνικέ διοικήσει, τον τομέα τη ελεία, την επιστημονική κοινότητα και μη κυβερνητικέ οργανώσει, όπω αποφασίσαν οι συντονιστέ, εκπροσωπούμεθα εμεί από την κυρία Πατράου Νέβε, την εισηγήτρια για την Πράσινη Βίβλο. Η δεύτερη συνάντηση αυτής της εβδομάδας είναι άτυπη συνάντηση των Υπουργών Αλίας 4 και 5 Μαΐου στο Βίγκο που συγκάλεσε η κυρία Σπινόζα η προεδρεύουσα, για να συζητηθεί η συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για την ε, μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής και την εξωτερική διάσταση πολιτικής. Σύμφωνα με την ε, διαθεσμική παράδοση που θεσπίστηκε από την Πρωτογαλλική Προεδρία του 2007, η πρόεδρος Επιτροπής μας, κυρία Φράγκα, κλήθηκε να συμμετάσχει σε αυτήν την συνάντηση και να λάβει μέρος συζήτηση με τους υπουργούς και τον υπατεπόση. Αναμφίβολα και η κυρία Πατραονέβες και η κυρία Φράγκο με ευχαρίστηση θα αναφέρουν τα αποτελέσματα των συνδύσεων του συνεδρίου στην επόμενη συνεδρία στις 2 Ιουνίου. Παίρνουμε τώρα σημείο 4 της ημερήσιας έταξης ψηφοφορία. Νέα όθηση στη στρατηγική τη βιώσιμη ανάπτυξη ευρωπαϊκή Υδατοκαλλιέργεια. Τον Απρίλιο η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση για την κοινοτική στρατηγική για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα υφόρο μέλλον για την ε, υδατοκαλλιέργεια, μια νέα όθηση για την στρατηγική για την υφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργεια. Έχουμε έκθεση πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου Γκέτο Μιλάνα από τους σοσιαλιστές. Μετά παρουσίαση του πρώτου γράφου εργασίας το Δεκέμβριο συζητήθηκε το θέμα αυτό πολλές συνεδρίες. Είχαμε και για την βιώσιμη δατοκαδιάθεση στις 23 Φεβρουαρίου δημόσια κρόση. Στην τελευταία συνεδρία στις 7 Απριλίου ο κύριος Μιλάνα παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης. Θεσπίσαμε ως προθεσμία κατάθεση τροπολιών την 13 Απριλίου. Λάβαμε 143 τροπολογίες που κατατέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή ΕΝΒΙ επίσης έστειλε την δική της γνωμοδότηση. Μεταξύ των πολιτικών ομάδων έχουμε και διάφορε συμβαστικέ τροπολογίε που κατέθηκαν τι πολιτικέ ομάδε. Πριν να περάσουμε στην ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μιλάνα, εάν θέλει να κάνει κάποιε διευκρινήσει όσον αφορά τον κατάλογο ψηφοφοριών. Κύριε Μιλάνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους. Προσπάθησα να συζητήσω τις ημέρες αυτές και εγώ ή οι συνεργάτες μου με τους συναδέλφους και τους συντονιστές σου, ώστε το κείμενο αυτό να είναι όσο πιο αποδεκτό γίνεται και προσπάθησα να καλύψω με θετικό τρόπο όλες τις τροπολογίες που είχαν εμφανιστεί συζήτηση των προηγούμενων συνεδριάσεων και να δεχθώ κατά, βάση, κατά συνέπεια στα όρια του maximum της έκθεσης κάποιες αλλαγές. Εγώ προσπάθησα να τις δεχτώ βεβαίως η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει τις θέσεις μας αλλά πιστέψτε με το έκανα με αίσθημα ευθύνης. Συχνά με περιορίζει το μέγεθος της έκθεσης ή ζητήματα που δεν θα μπορούσαν να υπαχθούν σε ένα από τα τέσσερα μεγάλα κεφάλαια της έκθεσης. Επαναλαμβάνω. Τα αιτήματα, ε, τα, τα, μεγάλα βασικά στοιχεία είναι πρώτον ενιαίος κανονισμός, ένας ενιαίος κανονισμός, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καλύπτει όλη την υδατοκαλλιέργεια εξ αρχή, αλλά σταδιακά να κάνει πιο οθολογική την νομοθετική αντιμετώπιση της υδατοκαλλιέργειας που αυτή τη στιγμή ε, εμφανίζονται σε πολλά νομικά κείμενα. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα πρέπει να, στο οποίο πρέπει να θεμελιώνει το κανονισμός είναι ένα σημαντικό ρυθμιστικό πλαίσιο, αυτό που λέμε ρυθμιστικό πλαίσιο της θάλασσας όπως το αποκαλούμε, μια έκφραση που θέλει να καλύψει μια να, να, να σημάνει μια ενοποιημένη αντιμετώπιση και πολιτική των ακτών που καλύπτει αλληλεία, υδατοκαλλιέργεια, τουρισμό, οικονομικές δραστηριότητες των θαλασσών και των εσωτερικών υδάτων. Τρίτη βασική, τρίτο βασικό στοιχείο, αύξηση της ε, ποιότητας, βελτίωση της ποιότητας. Άρα ανάγκη προστασίας της υγείας των καταναλωτών από τη μια πλευρά, της ευεξίας των ζώων από την άλλη, αλλά να αποτελέσει ένα συν στην ελληνική υδατοκαλλιέργεια. Άρα Τούτο πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο ως ένα στοιχείο βασικό της πολιτικής μας για τη θάλασσα. Ό,τι υπάγεται στη φιλοσοφία αυτή, όποια τροπολογία υπάγεται στη φιλοσοφία αυτή έγινε δεκτή από πλευρά μου. Ό,τι μπορούσε να υπονομεύσει κατά κάποιο τρόπο την θέση απορρίφθηκε. Παρά, διότι στις συζητήσεις των τελευταίων ε, μηνών, όσες φορές το συζητήσαμε το θέμα, τα ζητήματα αυτά, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ζητήματα που μας έβρισκαν όλους σύμφωνους. Μία τελική παρατήρηση για την θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος μας έστειλε μια σειρά συστάσεων. Είδατε στον κατάλογο ψηφοφορίας τις απόψεις μου για τον κατάλογο αυτό. Μη φοβάστε τα πλήν. Τα πλήν δεν είναι κρίση επί της ουσίας των θέσεων, είναι διότι στην έκθεση με άλλους όρους, όχι με τους ίδιους, αλλά οι θέσεις που προβλέπει η Επιτροπή, που προτείνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, βρίσκονται είτε στην αιτιολογική σκέψη, στις αιτιολογικές σκέψεις, είτε στις παραγράφους της εκθέσεως. Υπάρχει λοιπόν μία ουσιαστική συμφωνία των θέσεων της Επιτροπής ΕΜΒΗ με την δική σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί πραγματικά δουλέψατε πολύ καλά αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι υπήρχε μια αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των μεν από τους δε. Εγώ ξέρετε είμαι καινούριο βουλευτής και θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το θετικό πνεύμα, διότι η συνεργασία με όλους όσοι ε, δούλεψαν για την έκθεση αυτή ε, απαιτέλεσε για μένα πηγή πνευματικού πλούτου και ευκαιρία καλύτερης δουλειάς και βελτίωση της συνεργασίας μου. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Thank you very Ευχαριστώ κύριε Μαλάνα και ευχαριστώ και για τη σκληρή δουλειά που έχετε κάνει για την έκθεση. Να προχωρήσουμε. Έχετε όλη την κάρτα σας. Ξεκινούμε. 44 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό. Δεκτή τροπολογία ομόφωνα. 46. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Χωρίς την λέξη will. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Δεκτή. 11 υπέρ 9 κατά. Δεύτερο τμήμα. Η λέξη θα. Will. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Προτείνω από την 45 έως την 52 να ψηφίσουμε αν μπλοκ. Συμφωνείτε όλοι? Όχι, δεν συμφωνούν κάποιοι, άρα θα κάνουμε κάθε μία χωριστά. 45, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 47, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας Δεκτή. 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 49. Άρχεται. Ψηφίσατε. Πέρας. Δεκτή. 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Δεκ... Πέρας. Δεκτή. 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Καταπίπτει 53. 54 χωριστή ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 55. Όσο χωρίς κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό το τμήμα αυτό. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Τροπολογία 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 56 αποσύρεται. 57 είναι γλωσσική τροποποίηση. Άρα δεν ψηφίζουμε. 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζεται όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 66. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μια ψήφο. 65 είναι γλωσσική και πάλι ψηφίζουμε. Η 68 έχει αποσυρθεί. 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορία. Δεκτή. 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Δεκτή. 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 73 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Δεκτό το τμήμα αυτό. 74 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό. Πρώτη συμβαστική τροπολογία για την παράγραφο 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Οι 75, οι 76, οι 77, οι 78, οι 79 καταπίπτουν. 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέραση ψηφοφορία. Δεκτή. Η 81 έχει ε, αποσυρθεί. Η 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορία. Δεκτή. Συμβιβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζετε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Δεκτή. Η 84 καταπίπτει και η 85 και η 86 η 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρασε ψηφοφορία Δεκτή. 92. Καταπίπτει. 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή με μία ψήφο. Διαφορά. Η 89 αποσύρθηκε σήμερα το πρωί. 90 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό το κείμενο. 93 εδώ υπάρχει μια προφορική τροπολογία του κύριου Τσουκαλά. Θέλετε να, κάνετε, να παρουσιάσετε την προφορική σας τροπολογία? Α, την έχουμε στο τοσχέ μας. Σας ικανοποιεί? Ωραία, ευχαριστώ. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία του κύριου Τσουκαλά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Προχωρούμε. 94 η οποία καταπίπτει. 95-96 καταπίπτουν. 97 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 99 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή επίσης. 98 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 100 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσετε όλοι πέρας ψηφοφορίας δεκτή 101 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσετε πέρας ψηφοφορίας δεκτή 102 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσετε πέρας ψηφοφορίας επίσης δεκτή 103 αποσύρεται. 104 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 105 ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 107 άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Καταπίπτει, διορθώνει ο πρόεδρος. Και η 106 καταπίπτει. 108. Ψηφίζουμε την 108 άρχητη ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 110. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφίσετε Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 111 έχει αποσυρθεί. 112 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 113 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορία. δεκτή. 114 έχει αποσυρθεί. 115 ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 116 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας δεκτή. Με μικρή διαφορά. 117 τροπολογία έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας δεκτή. 118 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 119 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 120. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Επόμενη συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Άρα 123 τώρα. Όχι. Όχι. Καταπίπτει 123. Γυρίζουμε σελίδα. 129. Άρχεται η ψηφοφορία για την 129. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 130. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Κατερι... Απερίφθη το 131 μέχρι το 140 θα έλεγα να ψηφιστεί σε μία φορά, αλλά αφού υπάρχει αντίρρηση ε, θα ψηφίζεται κάθε τροπολογία χωριστά. 131. Ξεκινά ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Και εγκρίνεται. 132. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία Εγκρίνεται 133. Ξεκινάει η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 134. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 135. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 136. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. 137. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. 138. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 139. Ξεκινά. Το 140 ε, λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται 141 ψηφίσατε όλοι 142, Ψηφίσατε λίγοι. Εγκρίνεται. 143 ψηφίσατε όλοι λίγοι εγκρίνεται μετά προχωρούμε στα εκτιμώντας ε, ψηφίσατε λίγη ψηφοφορία και ε, απερίφθη. Δεύτερη τροπολογία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας ε, τροπολογία 4 αρχίζει, τελειώνει, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 και 6 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι, εγκρίνεται. 7. Ξεκινά. Λίγοι. Εδώ όμως έχουμε 10 υπέρ 10 κατά οπότε ε, καταπίπτει. Τροπολογία 8. Λίγη. Εγκρίνεται. 9. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Απορρίπτεται. 10. Ψηφίσατε. λίγοι. 11. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Εγκρίνεται. Μετά έχουμε τη συμβιβαστική τροπολογία 4. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 ε, ε, διαγράφεται, 13 διαγράφεται, 14 ε, ψηφίζεται. Λίγη. Και ε, εγκρίθηκε. 15. Ψηφίστε όλοι. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται 17. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Η 18 είναι γλωσσική. Η 19 ε, ε, απορρίπτεται η 5 ξεκινά εγκρίθηκε 20 καταπίπτει 21 και 22 είναι ταυτόσιμες ξεκινά Ψηφίσατε όλοι, λίγοι, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Ψηφίσατε όλοι, ε, λίγοι, εγκρίνεται. Η 23 τώρα. Καταπίπτει και 24 καταπίπτει, 25 ξεκινά ψηφοφορία. Λίγη, εγκρίθηκε, 26. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίθηκε. 27. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίθηκε. Γλωσσική 28 και 29. Προχωράμε στο 30. Ε, ψηφίσατε. Λίγη εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 7. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίθηκε. «31 μέχρι 34 διαγράφεται, προχωράμε στην 35, ξεκινάει η ψηφοφορία». Ψηφίσατε όλοι, ε, λίγοι και απερίφθη. 36 ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι και ε, με μία ψήφο εγκρίθηκε. 37. Ψήφισατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε 38. Υπέρ. Ε, Λίγοι. απορρίπτεται 39 λίγη εγκρίνεται 40 λίγη εγκρίνεται 41 καταπίπτει προχωράμε 42 η οποία είναι ε, χωριστή. Ξεκινά. Ε, ξεκινά η ψηφοφορία. Βλέπω ότι δεν ψηφίσαν όλοι. Είναι στο πρώτο μέρος του 42. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Το δεύτερο μέρος ε, ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Αποερίφθηκε. 43. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Εγκρίθηκε. Μετά, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ε, πρώτο εκτιμώντας ε, ξεκινά ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίθηκε. Δεύτερο εκτιμώντας. Ψηφίσατε όλοι. Τρίτο. Λίγοι απερίφθη δέλτα ξεκινά λίγη απερίφθη ε ξεκινά η ψηφοφορία λίγη εγκρίθηκε F ξεκινά λίγη ε, απερίφθη G ξεκινά λίγη ε, απερίφθη παράγραφος 1 λίγη απερίφθη 2 απερίφθη 3 λίγη απερίφθη 4 λίγη απερίφθη 5 απερίφθη 6 εγκρίνεται 7 απερίφθη 8 εγκρίνεται 9 Λίγη. Απερίευτη. 10. Εγκρίνεται. Ε, λίγη. Εγκρίθηκε. 11. Λίγη. Απερίφθη. 12. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Απερίφθη. 13. Απερίφθη. Και ε, ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα όπως ε, έχει τροποποιηθεί. Ψηφίσατε όλοι. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει, ε, τώρα ψήφισε. Λίγοι. Και εγκρίθηκε ομόφωνα. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μιλάνα, ο οποίος έκανε πολύ σωστή δουλειά με την ομόφωνη στήριξη όλων. Οπότε σας ευχαριστώ για αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή, ε, σας. υπομονή Νόμιζα ότι οι ψηφοφορίες θα κρατούσαν περισσότερη ώρα και χαίρομαι που τελειώσαμε τόσο γρήγορα. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στο 5 της ημερησίας διατάξεως, δηλαδή το καθεστώς εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αλληλείας και Ιδατοκαλλιέργειας στην προοπτική της μελλοντική μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ο εισηγητής είναι ο Αλάν Καντέκ αυτή η έκθεση κατά πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτάθηκε από το ΕΛΚ και ανελήφθη από τον Μισελ Καντέκ. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας έγινε στις 28 Ιανουαρίου. 26 Μαρτίου ο κύριος Καντέκ παρουσίασε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο προκάλεσε έντονες συζητήσεις μεταξύ των Ευρωβουλευτών και των εκπροσώπων της Γενικής Διευθύνσεως Μάρε και Εμπορίου σε αυτή την Επιτροπή. Πολλά θέματα ξανασυζητήθηκαν στην ακρόαση 8η Απριλίου σχετικά με την οργάνωση αγοράς και την αναθεώρηση της ΚΑΠ και τώρα ο κύριος Καντέκ θα παρουσιάσει την έκθεσή του και θα δώσω το λόγο στη συνέχεια και στους ευρωβουλευτές και στους εκπροσώπους της Επιτροπής. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Καντέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες υπενθυμίσεις, διότι εφ' εξής, αγαπητοί συνάδελφοι, ούτως ή άλλως απευθύνομαι και ευχαριστώ σε αυτούς που έχουν παραμείνει στην αίθουσα. Πάντα λέμε ότι οι καλύτεροι παραμένουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είστε οι καλύτεροι. Ούτω ή άλλω πρέπει να πω το εξή. Η έκθεση αυτή για τη καθεστώ εισαγωγή προϊόντων Αλλία και υδατοκατηλιέργεια είναι μετά από διαβουλεύσεις με εσά, με την διανομή και με τους όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο, αποτέλεσμα πολλών μηνών εργασίας. Έγινε η πρώτη παρουσίαση 16 Μαρτίου, έλαβα υπόψη τα διάφορα στοιχεία και πληροφορίες και επιχειρήματα μετά από την ακρόαση που είχαμε στις 8 Απριλίου για την οργάνωση της αγοράς. Είναι πρωταρχική σημασία να λάβει υπόψη αυτά στοιχεία τα οποία συμπεριλάβουν την εκθεσή μου. Απλώ έκανα κάποιες διαφορές, κάποιες συμπληρώσει μετά από τα σχάλια που έγιναν για να μπορέσω να παρουσιάσω με δομημένο τρόπο όλα τα στοιχεία που εξηγήθηκαν. Όπω εξηγείται και στην ετολική έκθεση, οργανώνεται η έκθεση γύρω από τέσσερι σειρέ ερωτήσεων. Πρώτα απ' όλα, τι ερωτήσει που αφορούν την κοινή εμπορική πολιτική, έτσι όπω εφαρμόστηκε μέχρι τώρα ε, για τα προϊόντα υδατοκαλλιεργία και καλλιέργεια, την συνεκτικότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη και υπεύθυνη αλία. Πράγμα που μα αφορά όλου. Δεύτερον, υπάρχει το θεμελιώδε θέμα των ε, προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και σε μεγαλύτερε ποσότητε ανταποκρίνονται στι απαιτήσει με αυτέ οι οποίε επιβάλλονται και στην Ευρωπαϊκή Αλία όσον αφορά το περιβάλλον, τα υγειονομικά θέματα, τα θέματα ποιότητα και τα κοινωνικά. Τρίτον, το θέμα Τη ε, επίγουσας μεταρρύθμισης κοινή αγορά εργασία στον τομέα τη αλληλεία και ιδιωτοκαλλιέργειας, στον οποίο οι κανονισμοί δεν φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, λαμβάνοντα υπόψη τους νέους ε, τελωνιακέ ε, αποβετήσεις μεταξύ άλλων. Και τέταρτο σημείο, το θέμα της ενημέρωσης του κατανοητή που κατά την άποψή μου είναι σημασία και η δημιουργία τελικά μιας πραγματικής ε, οικολογικής ετικέτας, ευρωπαϊκής οικολογικής ετικέτας για αυτά τα εισαγόμενα προϊόντα. Επίσης έκανε και κάτες παρατηρήσεις συμπληρωματικές για την υδατοκατέλγεια ε, αναφερόμενους στις ανταλλαγές απόψεων που είχαμε τον συνάδελφο Μιλάνα και με την κυρία Ράινες. Τα κύρια συμπεράσματα και οι συστάσεις τα εξής η πολιτική συστηματικού ανοίγματο στην οποία σε θέματα προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και αλίας ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεκτική με τα περιορισμούς οι οποίοι τίθενται όλο και περισσότερο για την κοινοτική αλία. Πρόκειται για δύο αντιφατικά πράγματα. Δεδομένου ότι καταλήγουμε στην αντιφατική κατάσταση και την παράδοξη κατάσταση που είναι απαράδεκτη και είναι η εξή. Πρώτα απ' όλα, για τη δική μα αλία ε, Υπάρχουν απαιτήσει ποιότητα, αλλά για να επιβιώσει η ευρωπαϊκή αλία οι τιμές δεν είναι επαρκείς. Υπάρχει λοιπόν κάτι το παράλογο εγώ. Τώρα, Δεδομένου ότι όλο και περισσότερο ανταγωνισμό υπάρχει από τα εισαγόμενα προϊόντα, βαχρυπρόθεσμα ίσω θυσιάσουμε την κοινοτική αλληλεία, διότι είμαστε υπέρ ε, της ε, απελευθέρωσης. Υπάρχουν διαφορετικά ε, οράματα για τους μεν και τους δε, αλλά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο όλοι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εξαρτώμεθα από την εισαγωγή πρώτων υλών από τις τρίτες χώρες το βλέπουμε αυτό για τα μεταποιημένα προϊόντα, κυρίως για τα προϊόντα τόνου και κυρίως στα πλαίσια των διαφόρων συμβάσεων οι οποίες έχουν ήδη συναυθεί ή είναι υποδιαπραγμάτευση. Αν δούμε προσεκτικά ποιε είναι αυτές, πώς ε, οι διαπραγματευσει εξελίσσονται, ε, θα δούμε ότι ο μεγαλυτερο κινδυνο είναι η διαπραγμάτευση άμυνα που γίνεται στα πλαίσια τη Πόλη. Η διαπραγμάτευση άμυνα λοιπόν θα καταλήξει ενδεχομένως στην ε, δραστική μείωση της ε, προστασίας τελωνιακής που επιβάλλεται στον τομέα αυτό για τα ε, μεταποιημένα και τα νοπά προϊόντα. Εκτός εάν σε τέτοιου είδου θέματα τελωνιακά εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω κάποια πράγματα ή κάτι μου διαφεύγει. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτός ο γύρος άρχισε το 2001, έπρεπε να διαρκέσει τρία χρόνια και είμαστε ήδη το 2010. Είναι λοιπόν ε, ίσως εύκολο να ανατρέψουμε τα πράγματα εάν θεωρήσουμε ότι τα τα προϊόντα το και αλίας είναι ευάλωτα και ευαίσθητα προϊόντα και τα αφαιρέσουμε από τι διαπραγματεύσει αυτέ που γίνονται στο γύρο της Δόχα. Πιστεύω ότι η ελβετική φόρμουλα είναι κάτι το οποίο μειώνει στο, ή μηδενίζει την ε, τελωνιακή προστασία για τα προϊόντα μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω αν ξέρετε όλοι την ελβετική φόρμουλα, θα σας την εξηγήσω για να χαλαρώσουμε. Δεδομένου ότι όλοι δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Είναι απλή η ελβετική φόρμουλα, πολύ απλή. Νέα δικαιώματα ίσον, ισούνται με τα παλιά συν συντελεστή, επί συντελεστή αυθαίρετο και κάτι άλλες αλχημίες, πράγματα που μας οδηγούν σε αφαίρετα αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω σε αμφισβήτηση εκ ε, μέρους εξονόματος όλων σας αυτή την αρχή. Το θέμα λοιπόν των προτιμήσεων ε, που χορηγούνται στους ε, διάφορους εταίρους με την εφαρμογή των κανόνων προέλευσης ίσως γίνει δευτερεύουσα σημασίας και οι μηχανισμοί που προβλέπει ο ΠΟΕ για να μπορέσουν τα διάφορα προϊόντα αλλιές και διατοκαλλιέργειας να φτάσει στις αγορές μας, φτάσει των αναγκών μας, είναι κάτι το οποίο θα είναι εντελώς απερχαιωμένο. Όλο και περισσότερο είναι απαιτητική η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τους ε, ε, δικούς της ε, τους αλλιείς, αλλά ενώ επιβάλλει για τα προϊόντα μας πολύ αυστηρούς κανόνες ποιότητας, για τις εισαγωγές δεν ε, επιμένει τόσο. Στις ε, ανταλλαγές απόψεων εγώ προσπάθησα όλα αυτά να τα τονίσω και να συμπεριλάβω όλα αυτά τα θέματα στην έκθεσή μου. Άκουσα τι είχατε να πείτε προσεκτικά. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την εφαρμογή των ίδιων κανόνων και των ίδιων απαιτήσεων για όλα τα προϊόντα, τα εισαγόμενα και τα δικά μας. Ε, δεδομένου όμως ότι κάποιες τρίτες χώρες έχουν μεγάλη πρόσβαση στις χώρες μας χωρίς όρους εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Υπό αυτές τις συνθήκες η λύση θα πρέπει να ανεβρεθεί με πολλαπλού τρόπου. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να εντείνουμε τη διεθνή συνεργασία σε θέματα αεφόρου διαχείριση των αποθεμάτων. Δεύτερον, να βοηθήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο τις χώρες που έχουν ανάγκη για να ε, πληρώσουν τα κριτήρια του Johannesburg. Να ανακληθούν ε, οι διάφορες ειδικέ προτιμήσεις οι οποίες έχουν δοθεί σε διάφορες χώρες σύμφωνα με του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Τρίτον, μεγάλη έλεγχη υγειονομική στις χώρες οι οποίες εισάγουν σε μας ήδη αλληλείας επιτόπου και στα ε, τελωνία. Και κυρίως αναφέρομαι στο παγκάσιο αυτό το στο ψάρι. Βεβαίως η έκθεση πρωτοβουλία η δική μου δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ όλο ιδιαίτερο με όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τις διαπραγματεύσει των πόρων. Δεν μπόρεσα να το εξετάσω αυτό το θέμα λεπτομεριακά. Την επόμενο χρόνο ξέρουμε όμως θα υποβάλουμε θετική πρόταση η Εκτελεστική Επιτροπή για μια νέα κοινή οργάνωση αγορά στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Νομίζω ότι αυτό είναι πρωταρχική σημασία. Διαπίστωσα στην έκθεσή μου ότι οι μηχανισμοί κοινή οργάνωση αγορά που υπενθυμίζω είναι σύστημα και ελάχιστες τιμές δεν επιτρέψουν στους αλλήλει μας να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερο ε, σε απαιτήσει υπάρχουν και όλο περισσότερα αλλιεύματα δικαιούνται να αλλιεύσουν. Το θέμα των εισαγωγών επίση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αναθεώρηση του συστήματο. Η Επιτροπή μα ότι είναι επίγον επίση να υπάρξει μια κοινοτική ε, οικολογική ετικέτα για να σταματήσει ο πολλαπλασιασμός, ο αυθαίρετος κατά κάποιο τρόπο, των ε, ιδιωτικών ετικετών. Είναι κάτι το οποίο το βρίσκει κανείς παντού και κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε από κοινοτικέ πλευρά. Ζητώ να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η μελέτη αυτή και νομίζω ότι είναι απαραίτητο και βεβαίως θέλω να διευκρινίσω ότι έχουν και κάποια αξία αυτέ οι ιδιωτικέ ετικέτε. Γιατί δεν υπήρχαν, θα ήταν τα πράγματα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ όλων των ετικετών που κυκλοφορούν. Νομίζω επίση ότι είναι απαραίτητο κάποιε παράγραφοι να ασχοληθούν με την όλη προβληματική τη αδετοκαλλιέργεια που ε, ε, εξηγούνται και στην έκθεση Μιλάνα, την οποία ψηφίσαμε ομόφωνα. Διότι νομίζω ότι είναι σημαντικά στον ε, όγκο των εισαγωμένων προϊόντων στον τομέα της αλίας στην κοινότητα. Υπάρχουν υποτρομές καθυστερήσεις σε αυτό τον τομέα. Πολλέ φορές συζητήσαμε και το είπα και στον πρόεδρο, ο Σολομός της Νορβηγίας και η Πόγκα από το Βιετνάμ είναι τα ε, κατεξοχήν ε, προϊόντα σε αυτό το τομέα. Στη συζήτηση 16 Μαρτίου Είπα ότι εάν θέλουμε να κάνουμε μια βιώσιμη κοινοτική ε, υδατοκαλλιέργεια θα επιτύχουμε μείωση των εισαγωγών παρεμφερών προϊόντων. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω σχόλια και παρατηρήσεις εκ μέρους σας, διότι αναμφίβολα θα τα υποβάλλετε. Με μεγάλη ευχαρίστηση συνεργαστώ μαζί σας και κυρίως με τους σκιώδεις εισηγητές για να βελτιωθεί και να συμπληρωθεί η έκθεσή μου. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι έχουμε και γνωμαδότηση εκ μέρους της συναδέλφου Ζανίκ Ζαντό, του συναδέλφου Γιάννικ Ζαντό, ο οποίος ναι. είναι από την Γιατί και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω διότι συνεργάστηκε ε, μαζί μου και για τη γνωμοδότηση αυτή. Πριν να καταθέσετε τροπολογίες, ο πρόεδρος θα σας πει ποιες είναι οι προθεσμίες, θα ήθελα να σας πω ότι διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά σφάλματα μετάφρασης γραπτής στην ε, αγγλική εκδοχή της έκθεσης και ίσως και σε άλλες γλωσσικές εκδοχές να υπάρχουν ε, ε, λάθη. Τα αγγλικά είναι μια γλώσσα που καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, εκτός από μένα φαίνεται. Τέλος πάντων, δεν είμαι και πολύ καλό στα αγγλικά. Ζήτησα λοιπόν στη γραμματεία να σας αποστείλει την διορθωμένη αγγλική εκδοχή της έκθεσης, πράγμα το οποίο έγινε χθε με mail και θα ήθελα στο του δυνατού να κάνετε τις επαληθεύσεις εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ του ε, γαλλικού εγγράφου του δικού μου και της αγγλικής μετάφρασης. Αυτά ήθελα να πω σύντομα κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι έχετε την έκθεση αυτή. Ήδη την ε, έχετε διαβάσει. Κύριε Πρόεδρε, σας, σας δίνω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ συνάδελφοι που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε κύριε Καντέκτη για την δουλειά σε μια πολύ σημαντική έκθεση. Συγχαρητήρια πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να πω κι εγώ δύο λόγια. Αναφέρεται ότι πραγματικά με τσαντίζει το θέμα του Παγκάσιος, όντως. Όσοι πήγατε στην έκθεση ε, προϊόντων της θαλάσσης την περασμένη εβδομάδα θα είδατε το περίπτερο του Βιετνάμ, το μεγαλύτερο περίπτερο όλων. Ε, ούτε σαν ποδοσφαιρικό γήπεδο ήταν με δεκάδες ε, Βιετναμέζους που υπέγραφαν ε, συμβόλαια για βουνά παγκάσιους από το δέλτα του Μεκόγκ. Υπέβαλα μια ερώτηση στην Επιτροπή και έλαβα απάντηση. Ε, τους ρώτησα πόσες επιθεωρήσεις έγιναν πέρυσι για υδατοκαλλιέργειας Παγκάσιους στο δέλτα του Μεκόγκ. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι τον περασμένο Οκτώβριο πήγαν δύο εξπέρ της Κομισιόν για δέκα μέρες και επισκέφθηκαν πέντε εργοστάσια μεταποίησης και τρία τρει χώρου υδατοκαλλιέργεια από τι 330 που έχουν άδεια να στέλνουν παγκάσιου στην Ένωση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αποδεκτό. Πριν από δύο χρόνια εισάγαμε 65.000 τόνους παγκάσιου στην Ένωση. Πέρσι, με βάση τα στοιχεία της απάντησης Επιτροπής, ο όγκος αυτός ήταν 220.000 τόνοι. Βουλιάζει η αγορά με αυτό το φτηνό ψάρι χαμηλής θρεπτικής ουσίας που περιέχει πολλά, πολλά ε, επικίνδυνα μηνοξέα και που δεν τηρεί και ε, που προέρχεται από ε, φάρμες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που ζητούν που ζητούν από τις δικές μας από τους δικούς μας χώρους υδατοκαλλιέργειας. Αν δείτε την ανάλυση και για τα ανοιχτή θαλάσσης ψάρια θα δείτε ότι, ο, ότι η δυνατότητα αυτή δεν είναι σωστή. Και ερώτησα την Επιτροπή γιατί έχουμε τόσο πολύ ψάρι κακής ποιότητας να μπαίνει στην αγορά, να καταστρέφει την αγορά, όχι μόνο για την υδατοκαλλιέργεια, αλλά και για την αλληλεία ανοιχτή θαλάσση. Γιατί δεν υπάρχει στο Βιετνάμ μόνιμη ομάδα επιθεωρητών που θα τους πληρώνουν οι Βιετναμέζοι. Αυτοί θέλουν πρόσβαση στην αγορά μας. Τέλο πάντων, τα έβγαλα από μέσα μου και ανοίγω τώρα τον λόγο για πολλούς ομιλητές, η κυρία Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κάντεκ, κατ' εμέ είναι ένα καλό και ισοσχελισμένο έγγραφο ε, έχουν περιληφθεί βασικά θέματα καταρχήν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνουμε ορισμένες απαιτήσει, να διατυπώσουμε απαιτήσει για τα προϊόντα εισαγωγής χρειαζόμαστε πληροφόρηση και θα πρέπει να προωθήσουμε και την αγορά μας υδατοκαλλιέργειες πρέπει να υπάρχει ισότητα ευκαιριών για τους εσωτερικούς παραγωγούς και αυτό είναι σημαντικό. Συμφωνούμε για το ελεύθερο εμπόριο αλλά θα πρέπει να, υπάρξουν, ε, ε, να υπάρξει σεβασμός και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των ευκαιριών και ε, δεν πρέπει ε, να υπάρχει μειονεκτική θέση ανταγωνιστική για τους δικούς μας παραγωγούς. Γενικώ όμως συγχαίρω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλέσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέκ για αυτή την έκθεση η οποία είναι πολύ σημαντική και η οποία αναφέρεται σε βασικά προβλήματα σχετικά με την αναθεώρηση της πολιτικής αλληλείας. Όντως υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για να ανοίξουμε την αγορά στα προϊόντα αυτά και να εξασφαλίσουμε την προσφορά αλλά η πλήρης απελευθέρωση μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά την αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εισαγωγέας ε, σε ολόκληρο ε, την Ιφίλιο και ε, πρέπει να φροντίσουμε η, η υδατοκαλλιέργεια της Πολωνίας να μην πληγεί όπως άλλωστε και η δατοκαλλιέργεια η ευρωπαϊκή από εισαγωγές. Ο κύριος Καντέκ αναφέρθηκε σε ένα πολύ βασικό θέμα, δηλαδή την έλλειψη ε, πληροφόρησης του καταναλωτού που θα πρέπει να έχει πολύ περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή του και ε, πολλές φορές οι καταναλωτές δεν έχουν καμία ενημέρωση σχετικά με την τιμή και ε, τα ψάρια τα οποία έχουν έχουν ε, ε, καλύτερη ε, διατροφική αξία και επικεντρώνονται στα φθηνά ψάρια. Πιστεύω όμως ότι αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αλλάξουν και μία συντονισμένη μέθοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο για τις ενδιαφερόμενες χώρες χρειάζεται. Ε- η έλλειψη συντονισμού οφείλεται εις ε, την ε, καθυστέρηση η οποία επιδεινώνει την θέση των Ευρωπαίων παραγωγών πράγμα το οποίο επαναλαμβάνουμε και συμφωνώ κύριε Πρόεδρε πρέπει οπωσδήποτε να καταρτιστούν λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι να γίνονται σεβαστοί και κανόνες οι οποίοι αναφέρουν αναφέρονται ή στους εξωτερικούς παραγωγούς όπως τους διαμέζους τους οποίους αναφέρατε. Ευχαριστώ κύριε Βαλέσα. Η κυρία Άντρες Μπερέα. Ευχαριστώ. Ξέρετε, ο κύριος Καντεκτού του ήδη τον συνεχάρει για την έκθεση και τις ε, παρεμβάσεις που είχαμε εδώ. Πρόκειται για μια έκθεση που καλύπτει πολλά θέματα που μας ενισχύουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να καταλάβουμε επίσης, να λάβουμε υπόψη και αυτό που προέκυψε και από την ακρόαση. Οι εισαγωγές είναι αναγκαίες. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη των εισαγωγών και εδώ είπε κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Βαλέντσα. Το θέμα του ελέγχου. Ο έλεγχος και από την άποψη της διατροφής, από την άποψη της διασφάλισης της ε, επισητιστικής υγεία, κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να προκύπτει στην επισήμανση, στο σήμα, τις απαιτήσει που θέλουμε να επιβάλλονται και δεύτερον το θέμα της πρόθεση στο εμπόριο. Το θέμα των εισαγωγών, το γεγονό ότι το ψάρι είναι ευαίσθητο προϊόν και πρέπει να απαιτείται η ίδια να επαντούνται οι ίδιε υποχρεώσει από τι τρίτε χώρε. Δεν πρέπει να συγχαίουμε το θέμα αυτό με τι διεθνεί συμφωνίε που έχουν δύο τμήματα. Ένα εμπορικό τμήμα και ένα τμήμα αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό αποτελεί υποχρέωση τη Ένωση. Πρέπει να διατηρήσουμε την διάσταση αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά η εμπορική διάσταση πρέπει να τηρείται μέσω τη εξειδίκευση των διεθνών συμφωνιών. Θεωρώ ότι το ζήτημα είναι να διευκρινίζουμε τι συνιστά έλεγχο, τι Ποιε είναι οι απαιτήσει κακού ανταγωνισμού που μπορεί να προκύψουν στι τρίτε αγορέ ει βάρο τη Ένωση. Ε, διευρύνοντας την αγορά, αν έχουμε μια, μια προσέγγιση αγορά-υγεία, έχουμε μια ισορροπία. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι χώρε αυτέ είναι εχθροί. Δεν θα λύσουμε έτσι την κατάσταση, αλλά λαμβάνοντα υπόψη αυτέ τι διαστάσει. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ο κύριο Γκάλαχαρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή. Εξαιρετική έκθεση. Πολύ σημαντική δουλειά έκανε για μας. Πολύ καλό το κείμενο. Συνεκτικό, πλήρες. Όχι μόνο για την Επιτροπή μας, αλλά και για τον κλάδο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι ενδιαφέρονται για το ζήτημα και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν καλές συστάσεις. Είναι σημαντικό να πρέπει και να μπορεί βεβαίως να κάνει επιθεωρήσεις στις ε, δομές υδατοκαλλιέργειες η Επιτροπή. Είναι σημαντικό να διεξάγονται αυτοί οι έλεγχοι συστηματικά, χωρίς προγενέστερη ενημέρωση ενδεχόμενα. Μπορεί αυτό να χρειάζεται να μπει στο πρωτόκολλο, αλλά θα μπορούσε να έχουμε μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση και να εξασφαλίζουμε ότι οι προδιαγραφές που ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα θα είναι του ιδίου επίπεδου με τις προδιαγραφές που θέτουμε στην εσωτερική αγορά. Όταν βλέπουμε τα εισαγόμενα προϊόντα ηλίας του 2007, είδαμε, βλέπουμε ότι εισήχθησαν 12 εκατομμύρια τόνοι, 55 δις ευρώ αξίας. Αυτό μας είπαν ότι αυξήθηκε με 10% χωρίς να λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό. Ε, θα φτάσει δηλαδή πάνω από τα 60 δις. Άρα μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Ούτως ή άλλως ωστόσο θα έπρεπε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των, δομών υδατοκαλλιέργειας διότι πρέπει να τους προσφέρουμε βιωσιμότητα και προγραμματισμό. Και αυτό που πλήττει τον ε, κλάδο περισσότερο είναι η γραφειοκρατία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε υψηλά στάνταρτ και να μην έχουμε τη γραφειοκρατία. Ας στείλουμε λοιπόν ένα σαφές μήνυμα, όχι μόνο στην Επιτροπή, η Επιτροπή δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα, αλλά και στα κράτη-μέλη. Και ιδίω διότι διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος από όταν επινοείται μία ιδέα μέχρι ότου να υπάρξει η ε, περιβαλλοντολογική μελέτη, οι δοκιμές και όλα αυτά χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί περισσότερο στην υδατοκαλλιέργεια διότι υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχει πίεση και και όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν ε, να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιήσουν τις ε, ευκαιρίες απασχόλησης. Ε, το έχω πει επανειλημμένος, αλλά ενδεχομένως ο πρόεδρος της Επιτροπής ή κάποιος άλλος θα μπορούσε να επέμβει διότι δεν χρειάζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας να ηγείται των συζητήσεων ε, σε θέματα αλίας δεν ε, ε, τα θέματα της εμπορίας αλίας δεν είναι θέματα του Επιτρόπου Αλίας αλλά τα θέματα του Επιτρόπου εμπορίου και θα έπρεπε η Επιτροπή μας να επιμείνει να αλλάξει το ισχύον καθεστώς και να επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του θέματος. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέκ για την εξαιρετική έκθεση την οποία κατήρτισε Πιστεύω ότι εξυπηρέτησε την ε, ε, Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και ε, χάραξε ένα δρόμο για το μέλλον. Αλλά δεν πρόκειται να επιτύχουμε παρά μόνο εάν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μία έκθεση απλώς στα χαρτιά. Θέλουμε να μπορέσει να εφαρμοστεί και να αποσταλεί στους υπευθύνους για λήψη αποφάσεων κατά, το, τρόπον ώστε να εφαρμοστεί άμεσα και όχι κάποτε στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Γκάλαχερ, ο κύριος Κομπάτσε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με τους άλλους ομιλητές που έλαβαν θέση για το περιεχόμενο της έκθεσης Καντέκ. Πολλές φορές είχα υπογραμμίσει τη, σημασία της έκθεσης για την κοινή πολιτική αλίας. Οι Πολωνοί ψαράδες λένε ότι η πολιτική η σωστή πολιτική τιμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση των ποσοστώσεων. Η έκθεση αυτή είναι τμήμα της πράσινης βιβλού για την ανοικοδόμη, για την αναμόρφωση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ρωτώ λοιπόν, να, θα ήθελα να λάβετε υπόψη κάτι τέτοιο στη διαμόρφωση της ε, πολιτικής αλληλείας. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Γκάλαγκερ δεν θα έπρεπε η έκθεση αυτή να μπει στο αρχείο. Σε μια προγενέστερη συνάντηση, την περασμένη ή την προπερασμένη, δεν θυμάμαι, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου είπε με ειλικρινή τρόπο ότι η απελευθέρωση των τιμών δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάσταση απόψεων και θέσεων. Πόσες προσπάθειες, πόσες αναλύσεις πρέπει να κάνουμε για να έχουμε κατευθυντήρες γραμμές που θα, με τις οποίες θα συμφωνούν όλοι για να λέμε τι είναι προς το συμφέρον και τι όχι προς, και τι δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής έλίας Η Γενική Διεύθυνση δεν θα έπρεπε μήπως ε, ενθαρρύνει υπερβολικά ή ευνοεί υπερβολικά την αγορά της από Ανατολής εις βάρος της δικής μας. Η κυρία Λέβαν. Ευχαριστώ. Τον κύριο Καντέκ πραγματικά ανέλαβε σημαντική, έκανε σημαντική δουλειά με αυτή την μεγάλη και αξιόλογη έκθεση και είναι καλό το ότι ξεκινούμε προσεκτικά στις εργασίες μας κοιτάζοντας εξ αρχής τις ανάγκες της αγωγής της Ένωσης. Ο αντίκτυπος των αναγκών αυτών, όχι μόνο για την ευρωπαϊκή αλία, αλλά και για την τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της αλλιές στις χώρες εκείνες. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που θα έπρεπε να το προσέξουμε προσεκτικά και να έχουμε επίγνωση των ζητημάτων. Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες απαιτήσει για τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον και θέματα υγείας, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το δρόμο αυτό τώρα. Δεν θέλουμε να συμβάλλουμε στην αλίευση ή την βλάβη του περιβάλλοντος στις χώρες από όπου προέρχονται τα ψάρια. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε και τι, κάνουμε, τι κάνουν τα δικά μας, η δική μας τόλη στα διεθνή είδα τα βάση των αλληλευτικών συμφωνιών. Οι αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής, για παράδειγμα, ε, έχουν περιορισμούς εξαγωγών για λόγους υγιεινής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πηγαίνουμε λοιπόν στα ύδατά τους, αγοράζουμε αλλιευτικά δικαιώματα και φέρνουμε ψάρια από την περιοχή αυτή στην Ευρώπη απευθείας. Και αυτό στα πρόβλημα. Ιδίως όταν Θέλουμε ισότιμη αντιμετώπιση και καταπολέμηση της, του αθέμητου ανταγωνισμού. Οι Αφρικανοί ψαράδες δεν έχουν την υποδομή που έχουμε εμείς, δεν έχουν τις δυνατότητες ε, στην υδατοκαλλιέργεια που έχουμε εμείς. Όταν πηγαίνουμε εμείς και αγοράζουμε ε, αλληλευτικά δικαιώματα για τα δικά τους ύδατα, ε, δεν μπορούμε να το περάσουμε αυτό ελαφρά την καρδία. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην έκθεση οι συνέπειες είναι ότι η συμπεριφορά αυτή είναι εις βάρος των χωρών, των αναπτυσσόμενων χωρών. Αν θέλουν να μας αντιμετωπίσουν σοβαρά οι χώρες αυτές, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας. Επίσης, δίνουμε έμφαση σε ζητήματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παράνομη αλία και να εξασφαλίσουμε ότι όντως παρέχουμε εγγυήσει ότι τα ψάρια που έχονται στην Ένωση έχουν αλληλευθεί νομίμως. Δεν αρκεί να ζητούμε από τις αναπτυσσόμενες χώρες να σταματήσουν οι ίδιες την παράνομη αλληλεία. Η έκθεση πρέπει να υπογραμμίζει και το γεγονός ότι πρέπει να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειες αυτές με καλύτερους ελέγχους ανά τον κόσμο. Όχι μόνο εδώ, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς είμαστε η μεγαλύτερη αγορά εισαγωγική. Πρέπει να βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται και έξω από τα νερά μας, γιατί είμαστε μεγάλοι. Αν δεν το κάνουμε αυτό εμείς, δύσκολα θα μπορέσει να υπάρχει εξασφάλιση ότι τα εισαγόμενα ψάρια έχουν όντως αλλιευθεί Εγώ είμαι υπέρ του οικολογικού συστήματος και της ανιχνευσιμότητας. Κάτι ουσιαστικό. Πρέπει να ξέρουμε πού αλλιεύθηκε το ψάρι, από ποιον, πότε και υπό ποιε συνθήκες. Αυτό είναι αυτονόητο σε ότι όταν μιλάμε για αλλιεύση στην ανοιχτή θάλασσα. Όταν, παίρνεις, όταν αγοράζεις αυγά, το κουτί με τα αυγά λέει ποιο τα παρήγαγε, τι έτρωγαν τα οικότες, ε, ζούσαν, ε, ήταν ε, ελεύθερης βοσκής ή όχι, όταν παίρνουμε για τα αυγά, τις πληροφορίες αυτές τις έχουμε. Όταν πάμε στα ψάρια όμως, το μόνο που ξέρουμε είναι πού περίπου ε, το ψάρι με βάση τον δείκτη του ΦΑΟ. Τίποτα άλλο. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των ψαριών. Κύριε Καντέκ, όταν μιλάτε για ένα κοινό οικολογικό σήμα για την Ευρώπη, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηρή στα κριτήρια. Γενικά, όχι μόνο εδώ. Πρέπει να... Δεν πρέπει να μπερδεύουμε αυτό το ζήτημα με το περιβαλλοντικό σήμα. Θέλουμε υψηλέ προδιαγραφέ από τη μία μεριά για τα προϊόντα εξωτερική προέλευση και από την άλλη μεριά να ξέρουμε ότι κάποιοι παραγωγοί τηρούν την, ε, ε, τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος ή ευεξίας των ζώων. Αυτό το θέμα δεν πρέπει να το ξεχνάμε και είναι δύο ζητήματα, δεν είναι ένα. Ευχαριστώ κύριε Λεβέν. Κύριε Μιλάνα. Εντάχει. Και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Καντέκ για τη δουλειά που έκανε. Πιστεύω ότι βάσει και αυτών που έλεγε κυρία Λαβέν πριν από λίγο, πρέπει να σκεφτούμε τον τύπο αυτό το, το μόνο πράγμα που θέλω να προτείνω στην έκθεση τον τύπο, την τυπολογία των εισαγόμενων προϊόντων. Εμείς έχουμε μία βεβαιότητα ότι υπάρχουν 4.300.000 τόνοι προϊόντων που εισάγονται και είναι προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάνω από 4 εκατομμύρια τόνοι που εισάγονται και που δεν είναι ψάρια που έχουν αλλιευθεί αλλά ψάρια που έχουν παραχθεί όπου το καθεστώς ελέγχου μπορεί να, ο έλεγχος μάλλον μπορεί να γίνει χωρίς προβλήματα. Ξέρουμε πού παράγεται. Εγώ λοιπόν θα έλεγα να κοιτάξουμε όχι τους εξαγωγείς μόνο, αλλά και τους εισαγωγή στην Ένωση. Το θέμα δεν είναι μόνο σχέσεις με την τοπική παραγωγή, αλλά και με τον έλεγχο της ε, αλυσίδας τη στιγμή της εισόδου. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε υπερβολικούς ελέγχους στη χώρα παραγωγής ε, του προϊόντος, αλλά ίσως και στις χώρες που κάπως έτσι χαλαρά εισάγουν το προϊόν. Κατόπιν έχουμε το πρόβλημα του, των ψαριών ανοιχτή θάλασσα που, ψαρα, που, που ψαρεύονται. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δεχτούμε τους αριθμούς. Η συζήτηση για το αν ένα ψάρι που ψαρεύεται από ένα, από ένα ευρωπαϊκό σκάφος ε, στα διεθνή ύδατα είναι εισαγόμενο ή όχι προϊόν. Εγώ θα έλεγα, δεν με ενδιαφέρει αυτό, αν εισάγεται ή όχι. Αλλά με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το επίθετο που χορηγούμε στο ψάρι αυτό. Είναι εισαγόμενο ή ευρωπαϊκό ψάρι. Θέλω όμως να έχω τον ορισμό, τον καθορισμό των όγκων. Διότι και εδώ η πολιτική πρέπει να διαμορφώνεται με βάση το φαινόμενο. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια πολιτική βάση της αποκλειστικής εμπορικής λογικής προσφοράς και ζήτησης. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική που θα προστατεύει τον καταναλωτή, τον επιχειρηματία και θα στηρίζεται σε μια ανάλυση ε, λεπτομεριακή του πώς και πού φτάνουν στην Ευρώπη οι ροές, οι εμπορικές ροές αλίας. Και νομίζω ότι αυτό το σημείο θα έπρεπε να το δει καλύτερη η έκθεση. Τη σχέση στο εσωτερικό των αλλιευόμενων ε, ψαριών του πώς τα προϊόντα αυτά, πόσα προϊόντα έρχονται στην Ευρώπη μέσω συμφωνιών και πόσοι μέσω διαδικασίας εισαγωγών. Συμφωνώ επίσης και με την κυρία Λοεβίν για την παράνομη αλληλεία. Καλό είναι να τα δούμε. Ένα τελευταίο θέμα που θεωρώ, στο οποίο θεωρώ ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καντέκ, είναι το θέμα της ανιχνευσιμότητας που θα πρέπει να ενισχύεται από μια πολιτική δημόσιο, δημόσιας επισήμανσης. Στο εισαγόμενο προϊόν πρέπει ο έλεγχος του, του πολιτικού σήματος να είναι έλεγχος δημόσιος. Στην εσωτερική αγορά το σύστημα των σημάτων παίζει ρόλο, άρα και η αυτοπιστοποίηση είναι σημαντική. Αλλά σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές πρέπει να βρούμε μια απάντηση, ψήφισμα ή νομοθετική λειτουργία ή διοικητική διαδικασία που θα επιτρέπει το σήμα να λειτουργεί ως ένα εργαλείο που θα προσφέρει ποιότητα. Για κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να είναι εύκολο. Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας για παράδειγμα. Το προϊόν που εισάγεται από υδατοκαλλιέργεια έχουμε τα στοιχεία, τα ξέρουμε, το μεγαλύτερο τμήμα είναι αυτό του εισαγόμενου, των εισαγόμενων ψαριών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Μιλάν. Αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος για την ε, σημασία της ε, αλίας στην Ευρώπη θα ήθελα να πω ότι είδα ένα DVD που έκανε στην Σενεγάλη και στη Σιέρα Λεόνη μια μη κυβερνητική ε, οργάνωση που είπε ότι υπάρχουν αλλιευτικά σκάφη παράνομα από την Κορέα και τη Ρωσία που υπεραλλιεύουν τις ακτές και εξαντλούν τα αλλιεύματα. Και μετά πηγαίνουν στα Κανάρια τα δίδουν σε δικά μας αλλιευτικά σκάφη και έτσι όλα αυτά τα αλλιεύματα, τα παράνομα φτάνουν ως νόμιμα στις δικές μας αγορές. Και δεν σας μιλώ για τις συνθήκες υπό τις οποίες αλλιεύαν τα ψάρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επιλύσουμε Και ξέρω ότι η κυρία Δαμανάκη θέλει να κάνει κάτι για την βελτίωση της αλλίας στην κοινότητα. Τώρα, όπως είπε ο κύριος Γκάλεξ, ο Ρίτσι Φλίν είναι ε, του τομέα της στην Ιρλανδία. Μας είπε στην ακρόαση εδώ ότι πριν μπορέσει να αλλιεύσει ένας ηχθειοκαλλιεργητής κάτι, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπακούσει σε περίπου 400 κανονισμούς ε, όλων των ε, ενεχόμενων γενικών διευθύνσεων κανόνες τι οποίες έχουν ε, θεσπίσει όχι μόνο τα κοινοτικά όργανα αλλά και τα εθνικά όργανα. Πρόκειται για εφιάλτη και αν δείτε ότι μας πλημμυρίζουν ε, πραγματικά τρομερές ποσότητες ε, αλλιευμάτων και δούμε από την άλλη μεριά πόσο επαχθείς είναι όλοι οι κανόνες του δικούς μας αλλιείς, κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή τι θα κάνει. Διότι όπως μας είπε η, από τους περίπου 300 ηχθειοκαλλιεργητές στο Βιετνάμ στους οποίους θα ενδεχομένως μπορεί να έγινε μια επιθεώρηση μόνο οι τρεις ήταν σωστοί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαμότζη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέκ για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Επίκαιρη με βάση και τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Είναι, υπάρχουν ορισμένοι τομείς ε, για τους οποίους έχουμε διαφορετική άποψη αλλά ούτω ή άλλω το κείμενο είναι μια εξαιρετική συνεισφορά στη συζήτηση για τη μεταρρυθμίση και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να μην ενισχυθεί, δεν πρόκειται να μπει σε κανένα σιρτάρι ή σε κανένα ντουλάπι στο γραφείο μας. Θα την λάβουμε σίγουρα υπόψη. Το κείμενο σας προφανώς είναι σε προκαταρκτική φάση, μπορεί να υπάρξουν ε, αλλά ανεξάρτητα από αυτό πιστεύω ότι έχετε πετύχει κάτι πολύ θετικό ήδη από τώρα. Κάποιες από τις προτάσεις σας δημιούργησαν ενδιαφέρουσες συζητήσει και στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και στην Γενική Διεύθυνση Αλληλευτικής Πολιτικής ε, Συζητήσει οποίε οποίες και τα ιδιαίτερα γραφεία των επιτρόπων. Από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να σας πω ότι αντίθετα από αυτό που αναφέρετε στο σχέδιο έκθεσή σας, δεν απετέλεσε η Αλία ποτέ ένα διαπραγματευτικό εργαλείο της γενικής μας διεύθυνσης για να πάρουμε κάτι άλλο από τους εμπορικούς εταίρους. Πάντα καταλαβαίναμε και λαμβάναμε υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα, του τομέα. Η έκθεσή σας σίγουρα αυξάνει και βελτιώνει την ε, ορατότητα και επίγνωση του κειμένου και σίγουρα βοηθήσατε να σκεφτούν καινούργια πράγματα πολλοί συνάδελφοι της Επιτροπής. Ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε πολλές συζητήσεις σε διάφορα ιδιαίτερα γραφεία. Επιπλέον μπορέσετε να καλύψετε το, τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Όταν, ε, τώρα μπαίνοντας στην ουσία της έκθεσης, ήδη έγιναν ε, ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων. Είχαμε συζητήσεις και στο γραφείο σας, είχαμε και συζητήσεις σε διεθνή βήματα. Πάνω από εκατοντάδες ε, σελίδων γραπτών κειμένων έχουν καλυφθεί ε, για τη συζήτηση. Δεν ήταν μάταια για μένα. Η συζήτηση που έχουμε σήμερα ήταν ενδιαφέρουσα και βλέπω ότι τα περισσότερα σχόλια που ακούστηκαν εδώ αφορούν κάποια κρίσιμα ζητήματα. Βιωσιμότητα του τομέα της αλληλείας, στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. Ισότιμη αντιμετώπιση, θεμητός ανταγωνισμός, ρόλος των δασμών για το μέλλον του κλάδου. να απαντήσω και σε κάποια σχόλια. Τα θέματα ισοτιμής αντιμετώπισης βιωσιμότητας τα έχουμε εξηγήσει. Η πολιτική της Επιτροπής είναι να λαμβάνει υπόψη την, τον ειδικό χαρακτήρα του κλάδου, κάτι που το πιστεύουμε ότι έγινε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμφανίζονται αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου στις ε, συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις σε διμερές και σε πολυμερές επίπεδο. Προφανώς υπάρχουν ορισμένα όρια που μπορούμε να πετύχουμε στο εγχείρημα αυτό. Πιστεύουμε ωστόσο ότι κάναμε ό,τι μπορούμε το μέγιστο για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά το NAMA και τις συνεχιζόμενες ε, διαπραγματεύσεις, που είναι ένα βασικό ζήτημα για την εμπορική πολιτική του κλάδου, μπορώ να σας πω ότι αυτή η ελβετική φόρμουλα περικοπής δασμών μπορεί να οδηγήσει στην διαγραφή των δασμών ως πιθανών ε, Το θέμα είναι, μπορεί στη φάση αυτή, η φόρμουλα αυτή να ε, επιληθεί βάση του τμήματος ε, του πακέτου για την πρόσβαση των μη γεωργικών προϊόντων στην αγορά ή μήπως θα πρέπει να βγάλουμε τα προϊόντα λίας από το σύνολο του, NAMA, του πακέτου NAMA. δεδομένων των ειδικών χαρακτηριστικών του κλάδου. Οι διαπραγματεύσεις των ΠΟΕ και στο ΓΚΑΤ δείχνουν ότι η φυστάμενη δομή του τμήματος AG πάνε πολύ παλιά πίσω. Υπάρχουν 53 ε, μέλη με διαφορετικά συμφέροντα που μπορούμε να επιδιώξουμε. Επίσης, Ξέρετε ότι και η Ένωση θέλει να κρατήσει το πακέτο αυτό της πρόσβασης στην αγορά χωρίς να ε, το πειράξει για να μην δεν θέλει να βγάλει διάφορους κλάδους γιατί θα ανοίξει ε, μια κερκόπορτα για άλλα προϊόντα άλλων χωρών που μπορεί να έχουν ε, ενδιαφέρον ή συμφέρον για συγκεκριμένους κλάδους. Στη φάση αυτή λοιπόν καλύτερα είναι να κρατήσουμε τον υφιστάμενο το υφιστάμενο σύστημα να μην ανοίξουμε δηλαδή πόρτες που μπορεί να ε, δημιουργήσουν προβλήματα. Να έχουμε δηλαδή ένα σύνολο κανόνων που θα είναι οριζόντιοι. Μετά, την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Ήρθε, ακούσαμε το επιχείρημα που αφορούσε την πρόσφατη παρέμβαση του Επιτρόπου κυρίου Δεχούχτ για την αναμόρφωση των ε, συμφωνιών ε, ε, DTA, κανοντα προτείνοντας ένα είδος DTA light. Ήθελε να πει ότι η Ένωση Δεν, αυτό δεν είχε να κάνει με τις αλλαγές προτεραιότητας της Επιτροπής στο ΝΑΜΑ. Μην ξεχνάτε ότι η συμφωνία αυτή για, τα μη γεωργικά προϊόντα, για την πρόσβαση στην αγορά μη γεωργικών προϊόντων, το ΝΑΜΑ, ε, είχε καθυστερήσει λόγω κάποιων ε, ε, φιλοδοξιών των ΗΠΑ. Αυτές οι φιλοδοξίες ωστόσο δεν ήταν πάντα σύμβατες με τις δικές μας είναι προφανές ότι αυτό που, θέλει, θέλουν οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί αν δεν υπάρξει και κάποια, αντι, ε, και κάποια αντιπροσφορά προς τις αναπτυσσόμενες χώρε. Και στο τέλος τέλος οι όλες οι πραγματεύσεις έχουν μια βάση, ατζέντα, μια βάση αναπτυξιακής ατζέντας. Άρα στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις χώρες αυτές. να τονίσω τώρα ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε εδώ. Το θέμα των προδιαγραφών και της αξιοπιστίας των προϊόντων, ιδίως των εισαγόμενων προϊόντων στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Το θέμα του Παγκάσιους που έφυξε ο πρόεδρος και τις πρόσφατες ε, επισκέψεις των συναδέλφων από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας στο Βιετνάμ. Στη φάση αυτή, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η έλεγχη των συναδέλφων από τις αντίστοιχες γενικές διευθύνσεις προφανώς ήταν αντίστοιχες με τους κινδύνους που προκύπτουν από το, τον όγκο εισαγωγών παγκάσιος. Καταγράφουμε το σχόλιο σας ότι δεν θεωρείται πως η έλεγχη αυτή είναι επαρκής. Θα τα μεταβιβάσω στις αρμόδιες αρχές. Επίσης κάποιοι, ε, κάποια μέλη της Επιτροπής έκαναν κάποια σχόλια ότι η Κομισιόν έχει πολύ περίπλοκους κανόνες ε, λειτουργίας του κλάδου, αλλά μην ξεχνάτε ότι από την άλλη μεριά πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι οι κανόνες αυτοί τηρούνται και εφαρμόζονται. Και αυτό συνιστά ευθύνη των κρατών μελών που είναι υπεύθυνα για την διεξαγωγή των υγειονομικών ε, έλεγχων στην Ένωση. Ξέρετε ότι έχουμε ένα σύνθετο πλέγμα κανόνων. Κάποιοι εμπορικοί εταίροι μας κατηγορούν ότι στην ουσία παρεμποδίζουμε το εμπόριο με ε, το επικαλούμενοι υγειονομικά ζητήματα και ότι θέλουμε απλά να, μειώσουμε τις, ε, να περιορίσουμε τις εισαγωγές στην ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύουμε ότι τα σχόλια αυτά δεν είναι σωστά. Οι έλεγχοι πληρούν και εφαρμόζουν την νομοθεσία. Να σας τομνήσω και μια συνάντηση στη Μαδρίτη που έγινε πρόσφατα με εμπλεκόμενους φορείς όπου σχολιάστηκε από κάποιους ο κίνδυνος γεννήσει σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές. Δεν πρέπει να γνωρούμε ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να παίρνουν από τους υπεύθυνους πολιτικούς ε, μηνύματα που μπορεί να τους οδηγήσουν στην αντίληψη ότι ένα προϊόν είναι ανθυγιεινό ή επικίνδυνο, ε, το παγκάσιος ξέρω εγώ. Υπάρχει ένας κίνδυνος κάτι τέτοιο να επηρεάσει την αγορά. Μια τελευταία παρατήρηση από πλευράς μου για το θέμα της ευθύνης. Σημειώνουμε και τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλια των κύριων βουλευτών. για το ότι τα πρόστιμα πρέπει να τα επιβάλλει η Επιτροπή. Εμείς στην, διασυν, στην ε, συνεργασία είχαμε, πρόσφατα είχαμε παρουσιάσει τη θέση μας. Καμία, να τονίσω ότι καμία υπηρεσία της Επιτροπής δεν δρά μόνη της. Με μία φωνή μιλάει η Επιτροπή και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την αρχή της συλλογικότητας. Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρείτε την Α ή τη Β γενική διεύθυνση ένοχη για την Α ή Β πολιτική. Στις δε εμπορικέ διαπραγματεύσεις μην ξεχνάτε ότι η Επιτροπή βρά η υποστενή παρακολούθηση και σε πλήρη συνεργασία με τους διάφορους εμπλεκόμενους κλάδους. Οι διαπραγματευτικές οδηγίες μας υιοθετούνται από το Συμβούλιο, με τα κράτη-μέλη τακτικά, το ίδιο και το Κοινοβούλιο ιδίως μετά την θέση ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, η συνεργασία αυτή θα είναι στενότερη. Επίσης, έχουμε τακτικό και ζωντανό συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτές είναι οι πρώτες παρατηρήσεις μου για κάποια από τα βασικά θέματα. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Αλληλευτικής Πολιτικής θέλει να κάνει κάποια σχόλια για δικούς του τομείς αρμοδιότητες. Ο κύριος Ράμπο από την Επιτροπή. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα. Notre grand intérêt Επιτρέψτε μου να πω πόσο πολύ μας ενδιαφέρει η έκθεση αυτή, διότι όπως ελέγχθηκε την τελευταία φορά είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Φτάνει την κατάλληλη στιγμή, τη στιγμή την οποία θέλουμε να κάνουμε την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και κυρίως το θέμα της οργάνωσης της, αγοράς. Σε σχέση με το αρχικό έγγραφο εργασίας, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή βελτιώθηκε, ε, τροποποιήθηκε με βάση πληροφορίες οι οποίες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την συνέχεια της συζήτησης. Θα ήθελα να κάνω δύο εισαγωγικέ παρατηρήσεις και μετά να αρχίσω τις επί του θέματος παρατηρήσεις. Αυτή η έννοια συστηματικού ανήματος της κοινοτική αγοράς θα πρέπει να πω ότι έχει ως στόχο όχι μόνο να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών μας, αλλά να επιτρέψει να υπάρχει και στον ε, ε, τομέα της μεταποίησης των προϊόντων της αλίας ε, η δραστηριότητα. Θα πρέπει να δούμε το εξή. Οι επιπτώσει των εισαγωγών θα πρέπει να εκτιμώνται κατά περίπτωση. Δεδομένου κύριε Πρόεδρε ότι εσείς αναφέρετε το παγκάσιο και τις εισαγωγές, τις μεγάλες ποσότητες, τις τεράστιες ποσότητες σε παγκασίου, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό έχει άμεση επιπτώσεις επί του επίπεδου των τιμών. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε ανάγκες των καταναλωτών και να προσελκύσουμε με αυτό το ψάρι και νέους καταναλωτές οι οποίοι σήμερα όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε δεδομένου ότι διαπιστώνω αυτό δεν είναι το καλύτερο ψάρι του κόσμου κατευθύνονται σε άλλα ψάρια. Άρα μπορούμε και εδώ να δούμε κάτι το θετικό. Δεύτερο στοιχείο. Είμαστε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή αλλιευτικής ε, πολιτικής που είναι 36 τρόπου. Ο πρώτο είναι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα τη της κατά πρώτο λόγο της κοινοτική και βεβαίως της ε, παγκοσμίου δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σύνορα για τη δική μας αλληλεία και έχουμε αλληλευτικά σκάφη τα οποία αλλιεύουν και εκτός κοινοτικών υδάτων και έχουμε ισχυρή παρουσία. Δεύτερο στοιχείο. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει επίσης ως στόχο ίσως να απλοποιεί και αυτό είναι κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Γκάλαχης πόσο πολύπλοκο είναι να λιεύσει ένας ε, κοινοτικός αλλιές, πόσους κανονισμούς θα πρέπει να σεβαστεί. Στόχος μας λοιπόν είναι να βελτιώσουμε την διαχείριση της κοινοτικής αλίας και να απλουστεύσουμε τα πράγματα και βεβαίως κατά τρίτο λόγο να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και της αλληλευτικής βιομηχανίας και του αλληλευτικού μας στόλου σε σχέση με μια παγκοσμιοποιημένη αλληλευτική αγορά, όπως είπε και ο κύριος Καντέκ. Τώρα, μετά από αυτές τις αγωγικές παρατηρήσεις, θα ήθελα να κάνω πέντε παρατηρήσεις, τα οποία θεωρώ ότι αποτελούν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των αγορών της αλίας και της ιδιωτικατιέργειας ότι είναι σημεία, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν, να μελετηθούν, ώστε να οδηγηθούμε σε πιο υγιή και δίκαιο ανταγωνισμό. Ανέφερε ο συνάδελφός σας το σεμινάριο της Μαδρίτης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέκ, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το σεμινάριο, για τον υγιή ανταγωνισμό. τον οποίο μπορούμε βάσει πέντε στοιχείων να κάνουμε πιο δυναμικό. Το θέμα της υγείας, το υγειονομικό. Όπως είπε ο κ. Ζοκατέκη, πιστεύουμε ότι για θέματα ελέγχου, σε θέματα υγείας, για να προσφέρουμε τους καταναλωτές, έχουμε τον καλύτερο ε, μηχανισμό στον κόσμο. Αυτό είναι αναμφίβολο. Όπως αναφέρθηκα, Υπάρχουν κάποιε δυσκολίε που αντιμετωπίζουν κάποια εταίροι μα, κυρίω από τι αναπτυσσόμενε χώρε. Και πιστεύω ότι υπάρχουν μηχανισμοί αμοιβαία αρρωγή και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ που επιτρέπει στι αναπτυσσόμενε χώρε να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτό το καθεστώς. Επίση, θα ήθελα να αναφέρω ότι στα εκατομμύρια τόνους που εισάγουμε μέχρι αποδείξεις του εναντίου δεν είχαμε μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Και δεν θα πρέπει να επιμένουμε και σε χώρες ή σε ε, προϊόντα μόνο. Το ποσό, το, συγγνώμη, το, σε μεγαλύτερη ποσότητα από το εξωτερικό αυτό το οποίο εισάγουμε είναι γαρίδες. Και βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε και χωρίς τη συνδρομή της Νορβηγίας και της Ισλανδίας και ποτέ από τις δύο χώρες αυτές δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Τώρα, η ποιότητα. Στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση πρέπει να πω ότι έχει επιτευχθεί πρόεδρο εδώ και 10 χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο διαφοροποιεί τα κοινοτικά αλλιευτικά προϊόντα από τα άλλα που θα πρέπει να γίνουν μεγάλες προσπάθειες και στα πλαίσια της μεταρρύθμισης πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε και τα μέσα αλλά και τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε την ποιότητα των ευρωπαϊκών αλλιευτικών προϊόντων ώστε να έχουν καλύτερη θέση στην αγορά της μεταποίησης ή για άμεση κατανάλωση από τους Ευρωπαίους παρατήρηση σε σχέση με την ε, νυχνευσιμότητα. Καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι η μεταρρύθμιση του κανονισμού για τον έλεγχο που εγκρίθηκε πέρσι επέτρεψε για πρώτη φορά το θέμα της χνηλασιμότητας των αλληλευτικών προϊόντων να το επεκτείνουμε από το ε, από τον ηχθειοκαλλιεργητή, από το πλοίο εκεί που αλλιεύονται, μέχρι τον καταναλωτή. Η γλασιμότητα, λοιπόν που είχε τεθεί σε ισχύ το 2002 αρχίζει όπως σας λέγω ή από την φάρμα του ηχθειοκαλλιεργητή ή από το πλοίο. Από του χρόνου θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι και όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή εγκρίνουμε τα μέτρα και τους τρόπους με τους οποίους θα διευκολυνθεί η η γλασιμότητα για τα κράτη-μέλη. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν και ευθύνες για όλους τους εταίρους μας και πράγμα που θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερη πολιτική επικοινωνίας για τα αλλιευτικά προϊόντα προς όφελο των καταναλωτών. Όσον αφορά την UU, έγινε την προηγούμενη μέρα στο Buenos Aires μία συνάντηση, στην οποία συμμετείχαμε και πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλληλεία δεν θεωρείται ως εμπόδιο για την εμπόριο, αλλά πρωταρχικής σημασίας μέσων για την διαχείριση της παγκοσμιολίας. Υπάρχουν ακόμη δυσκολίες, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη χώρες που δεν μπορούν να δώσουν την πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι καλύπτονται οι εισαγωγές μας σε ποσοστό 100% από τα συστήματα πιστοποίησης αυτό είναι κάτι το οποίο μας το είπαν οι εταίροι και τέσσερις μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πρόκληση πραγματικά είναι μια πρόκληση στην οποία ανταποκριθήκαμε. Τώρα θα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση, στη φάση ελέγχου, όπως κάνουμε και στον τομέα των υγειονομών, ώστε να δούμε κατά πόσον οι αρχές που δίδουν αυτά τα πιστοποιητικά ότι είναι νόμιμη η αλία, ότι τα πλοία ενεργούν με νόμιμο τρόπο, το κάνουν σωστά. Και εδώ θα μας συνδράμει η σχετικός οργανισμός για τους ελέγχους. Τώρα, όσον αφορά τη σήμανση. Η σήμανση είναι πρωταρχική σημασία στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των αγορών των ληφτικών προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Σήμερα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το όλο σύστημα υποχρεωτικών πληροφοριών που θεωρούν όλοι ότι είναι ανεπαρκείς. Ε, ζώνες αλίευσης, ε, ζώνες άλλα στοιχεία και όνομα του ψαριού. Αυτό όλο το σύστημα θα ανεωρηθεί εκ βαθέων. Το άλλο θέμα είναι ότι θα και αυτό είναι μια άλλη ιδέα, είναι ότι θα πρέπει σε θελούσια βάση να δούμε πώς μπορούμε να πλαισιώσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και αναφέρομαι στην σήμανση και στις παρατηρήσεις που έγιναν όσον αφορά την οικολογική σήμανση, το eco-labeling για το δίκαιο εμπόριο Και βεβαίως μία από τι προκλήσει στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούμε στα πλαίσια μεταρρύθμιση της αγοράς εργασία είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την σωστή σήμανση στα ψάρια, ώστε όχι μόνο να έχουμε πιο ακριβείς προφορίες για τον καταναλωτή, αλλά να επιτρέψουμε οι προφορίες που εμπεριέχονται να είναι χρήσιμες. Αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε, για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Αντρές Περέα, θέλετε να αντιδράσετε. Δεν θέλω να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση, αλλά αν θέλετε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο. Όχι, μα δεν έχω κάτι τέτοιο σκοπό. Να παρακαλέσω τον κύριο Στίβενσον το εξή. Μιλήσατε, πρόεδρε, για την παράνομη αλία. Κάτι που μα ανησυχεί όλου. και τις περιπτώσεις διευκόλυνσης, ας πούμε, να, ε, μια περίπτωση κορεάτικα σκάφη που βγάζουν ψάρια στα Κανάρια. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα αντίγραφο τη, του, του, του, των πληροφοριών που λάβατε για να έχουμε μια εικό, εικόνα της κατάστασης. Θα σας στείλω ένα αντίγραφο των πληροφοριών. Ο κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή ήταν ε, πολύ πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας όλους και θα ε, απαριθμίσω ένα προς ένα τα θέματα ε, και θα σημειώνω παρατηρήσεις. Εσείς κύριε Πρόεδρε τονίσατε τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι σημαντικές εισαγωγές ε, παγκάσιου από το Βιετνάμ 220.000 ε, τόνοι το χρόνο για διατροφή μηδέν διατροφική αξία 0, 0 ε, ωμέγα 3 οπότε να μην μας λένε ανοησίες υπάρχουν ε, τέσσερις χιλιάδες υδατοκαλλιέργειες ε, στον Μεκόγκ οπότε με συγχωρείτε ε, αλλά τρεις έλεγχοι σε τέσσερις χιλιάδες σε 4.000 ε, ε, καλλιέργειες ε, στον Μεκόγκ που είναι ένα φοδευτικό σύστημα γεμάτο βακτηρίδια, μικρόβια, το ξέρουμε όλοι. Τρεις έλεγχοι το χρόνο δεν επαρκούν, μην μας λένε ανοησίες. Επίσης μιλήσαμε για ισότητα και ε, ε, ε, απελευθέρωση αλλά ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται συλλογικά όχι με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Βαλέσα τόνισε επίσης το θέμα της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με τις εισαγωγές ήταν σημαντικό το ξαναναφέραμε και κατάλαβα το μήνυμά σας ε, σχετικά με την ε, ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν είναι ασύμβατα αυτά και πρέπει να περιληφθούν επίσης στην έκθεση. Θα πρέπει να το αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα στην έκθεση. Ο φίλος μου, ο κύριος Γκάλαχερ, αναφέρθηκε για τις τις ε, ε, ε, υδατοκαλλιέργειες τρίτες χώρες τις οποίες δεν μπορούμε να, να ελέγξουμε με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Ένας άλλος συνάδελφος αναφέρθηκε στη θέση της Γενικής Διευθύνσεως Εμπορίου σε σχέση με άλλων ε, γενικών διευθύνσεων και συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπες. Όσον αφορά αναπτυξιακή βοήθεια, θα επεκταθώ στο θέμα αυτό αν θέλετε, ε, αλλά το θέμα δεν είναι ε, να τιμωρηθούν μέσω των ε, αποφάσεων που θα λάβουμε εμείς για να ενισχύσουμε ε, την ε, αλία μας. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Άλλωστε, όντως, πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα την παράνομη αλία και όσο για την ιχνηλασιμότητα θα πρέπει να υπάρχει ε, ποιοτικά, κοινοτικά, περιβαλλοντολογικά αυτή η ιχνηλασιμότητα. Όλοι συμφωνούμε. Ε, ε, σας είπα 250.000 τόνοι έρχονται από το Βιετνάμ και ακόμη περισσότεροι από άλλες τρίτες χώρες άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους των εισαγωγών. Ε, ευχαριστώ ε, για τα θετικά σχόλια που εξεφράστηκαν για σχετικά με την έκθεση αυτή και αν κατάλαβα καλά ε, νομίζω ότι όντως κατάλαβα το νόημα των παρατηρήσεων αποδέχεστε την έκθεσή μου, από την άλλη πλευρά όμως μου λέτε ότι πρέπει να είναι πιο απλοποιημένη. Ε, διότι εδώ μας λέγουν ότι είναι καλή η έκθεσή σας αλλά δεν πρόκειται να κινηθούμε ε, έτσι τουλάχιστον μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας βοηθήσουμε όμως ε, να κινηθείτε και θα σας βοηθήσουμε να κινήσετε και τον κύριο Ντεγκύρτ γι' αυτό και υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αδιαφυσβήτητα σχετικά με την έκθεση αυτή αλλά σιγά σιγά καταρχήν θέλω να σας ε, συγχαρώ για την παρέμβασή σας η οποία ήταν εξαιρετική και πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την έκθεση την οποία μας είχατε διαβάσει στην πρώτη παρέμβασή σας. Και όσον αφορά αυτή την παρέμβαση μας είπατε ότι ε, νέα προσέγγιση σχετικά με τα νάμας δεν θα είναι εύκολη, ε, θα υπάρξουν επιπτώσεις και σε άλλες χώρες, η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν ξέρουμε αν ο κύριος Ντεγκούρτ θέλει, να, θέλει να αλλάξει το πακέτο των ε, εμπορικών προσβάσεων ε, ουσιαστικά όμως αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ε, ότι θέλουμε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ε, ευρωπαϊκή αλληλεία και να προστατεύσουμε και τους συνεργάτες μας εμείς έχουμε την καλή θέληση και θέλουμε να επιτύχουμε και τίποτα δεν θα μας εμποδίσει. Αυτά είχα να σας πω εκ μέρους ε, σαν σχόλια προς τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ήδη έχουμε κάνει συζητήσεις, ε, θα ξαναέχουμε, αλλά ε, ελπίζω ότι καταλάβατε το μήνυμά μου και παρακαλώ να το μεταδώσετε. Όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση ε, νομίζω ότι υπήρξε ε, μία κίνηση ε, αλλά ελάχιστη μάλλον ακαμψία της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ και πολύ λυπούμε σας το λέω όπως το σκέφτομαι Κρισιό διότι εφόσον ο κύριος Σομογγί μας μίλησε ε, για ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής μας λυπεί διότι εγώ δεν θέλω να υπάρχει πόλεμος μεταξύ των επιτροπών. Μία είναι η επίτροπη, όλοι οι επίτροποι ε, μία είναι η επιτροπή όλοι οι επίτροποι είναι ίσοι ε, και ε, το, ενώ στο κοινοβούλιο έχουμε διαφορές απόψεων και ψηφίζουμε για να προωθήσουμε τα θέματα θα πρέπει και εσείς να μπορείτε να επιτύχετε. Όταν λοιπόν λέτε ότι δεν υπάρχει άμεση επίπτωση στις τιμές μέσω των εισαγωγών ε, δεν είναι αλήθεια γιατί αυτό είναι διαφυσβήτητο, είναι αριθμητική. Ε, συζήτησα με έναν παραγωγό παγκασίου κατά την έκθεση ΣΥΦΟΥ την περασμένη εβδομάδα με συγχωρείτε, πρόκειται για εισαγωγέα και όχι για παραγωγό και αν δείτε ε, ποια είναι η τιμή που παράγεται, η τιμή που εισάγεται και η τιμή που πωλείται υπάρχει επιρροή επί των τιμών. Δεν υπάρχει δηλαδή μία ίση και υγιής ε, κατάσταση ανταγωνισμού. Πιστεύω ότι υπάρχει ε, αθέμητος ανταγωνισμός και αυτό ήθελα να πω. Και τέλος καταλήγοντας Θα ήθελα να σας πω και σας το λέω κατευθείαν, αλλά καλό θα ήταν ίσως ε, να το επαναλάβω ότι σας καλώ να ε, μελετήσετε αν ως ε, ε, εκλεγμένοι υπεύθυνοι για λήψη αποφάσεων πολιτικών πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις προδιαγραφές γιατί όλα θα περιπλακούν ή αν είναι άκαπτε ε, οι επιταγές της πολιτικής αλληλείας και αν ε, δεν πρέπει να παρέμβουμε. Και εγώ ε, θα αρνηθώ να δεχτώ αυτή τη θέση. Πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβουμε για να βοηθήσουν και να σώσουμε την αλληλεία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Σίγουρα το θέμα αυτό πάντα ανάβει και τα μέλη της Επιτροπής και την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες στην έκθεση είναι 17 Μαΐου, Παρασκευή, 12 η ώρα, μεθαύριο δηλαδή. Τι θέλετε κύριε Λεβέν. Θα πρότεινα να παραταθεί η προθεσμία μέχρι την άλλη εβδομάδα. Υπάρχουν και τα μεταφραστικά προβλήματα στην έκθεση. Είναι σημαντική, πολύ σημαντική έκθεση. Θα ήθελα να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να το ξαναδιαβάσουμε. Θα πρότεινα να αναβάλουμε την προθεσμία την άλλη εβδομάδα. Είναι σημαντική έκθεση. Δεν το πολύ θέλω να σας πω την αλήθεια. Οι προθεσμίες έγιναν, ε, συμφωνήθηκαν με τους συντονιστές. Και γιατί είναι αυτό. Κανονικά θα ψηφίζαμε στις 2 Ιουνίου στην Επιτροπή. Άρα θα περνάγαμε στην Ολομέλεια του Ιουλίου, πριν τις διακοπές του καλοκαιριού. Ακούστε τη συζήτηση σήμερα το πρωί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να τηρηθούν ε, οι προθεσμίες και να έχετε τις προτοπολογίες μέχρι την Παρασκευή. Αλλιώ όμως υπάρχει κίνδυνος να αναβάλουμε την όλη την ψηφοφορία του Σεπτέμβριου. Για το... Είναι σημαντικό λοιπόν να περάσει πριν το καλοκαίρι η έκθεση. Τι λέτε κύριε Καντέκ. Νομίζω ότι αν θέλουμε να τηρήσουμε το timing πρέπει να το τηρήσουμε. Τι να σου πω, να βάλουμε κανένα δύο μέρες ακόμα. Τι να σας πω. Ορίστε. 11, τρίτη, τρίτη, τρίτη, επόμενη τρίτη, 11 του μηνός. Αν το επιτρέπετε πρόεδρε, 11 του μηνός οι συντονιστές συμφώνησαν όλες οι εκθέσεις που εξετάζουμε σήμερα να έχουν προθεσμία 12 το μεσημέρι της Παρασκευής. Αν ζητάτε αυτό θα έχουμε αιτήματα και για τα άλλα. Ανατρέπει το χρονοδιάγραμμα αυτό. Μα είναι ειδική περίπτωση αυτή. Υπάρχουν και τα γλωσσικά προβλήματα. Πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε. Πρόκειται για ειδική περίπτωση. Εντάξει. Εντάξει. Ελπίζω να συμφωνήσετε ότι αυτό δεν αποτελεί προηγούμενο για τις άλλες εκθέσεις. Με την έγκριση του εισηγητή η προθεσμία είναι πλέον τρίτη 12 η ώρα, η επόμενη τρίτη 12 η ώρα. Ελπίζω να μην ε, ανατρέψει όλο το χρονοδιάγραμμα. και ελπίζουμε να το ψηφίσουμε πάλι στις 2 Ιουνίου στην Επιτροπή και να πάει στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Λοιπόν, προχωρούμε. Το 6. Ο έλεγχος από τα κράτη-μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι η επί της ουσίας αρμόδια με βάση την κανονική νομοθετική διαδικασία με πρόταση επιτροπής για τον κανονισμό που καθορίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές για τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη-μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιότητων από την Επιτροπή. Η νομική επιτροπή ενέφησε την έκθεση στον Γιώζεφ Σάιερ. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή Αλίας και όλα τα άλλα και άλλες, άλλες νομοθετικές ε, αρμόδιες να ετοιμάσει μια έκθεση για αυτό το σημαντικό θέμα. Η ψηφοφορία στην Νομική Επιτροπή προβλέπεται για το τέλος Ιουνίου. Όσοι οι συντονιστές αποφάσισαν να δώσουν στον κύριο Κούν την οδηγία αυτή, την γνωμοδότηση αυτή, που είναι ο μόνιμος εισηγητής μας για θέματα επιτροπολογίας. Λόγω όμως του στενού χρονοδιαγράμματος, ο κύριος Κούν ετοίμασε ήδη ένα σχέδιο γνωμοδότησης, δεν μπορεί να έρθει και ζήτησε τον κύριο, από τον κύριο Καντέκ να παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καντέκ, να επαναλάβω. Για την έκθεση αυτή η προθεσμία είναι 12 η ώρα την Παρασκευή. Κύριε Καντέκ, έχετε το λόγο και εκ νέου. Καταρχά να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματο του συναδέλφου κύριου Κούν, που δεν μπορεί να έρθει. Έχει υποχρεώσεις ε, στην εκλογική του περιφέρεια. Μου ζήτησε λοιπόν να τον αντικαταστήσω και θα το προσπαθήσω. Να σα κάνω μια σύντομη παρουσίαση του θέματο που δεν την ξέρω καλά, θα το παρουσιάσω. Όπως ξέρετε, στην επόμενη Ολομέλεια το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την έκθεση Σάιερ για την... τις κατεξοδοτήσεις πράξης. Και η πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό που θέτει τους γενικούς κανόνες ε, για τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη-μέλη των ασκήσεων ε, των εκτελεστικών νομοθετήρων από την Επιτροπή, επί της οποίας μας ζήτησε να παρουσιάσουμε γνωμοδότηση η νομική επιτροπή, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συμπλήρωμα της προηγούμενης εκθέσης του κ. Ζάγερ για τις εκτελεστικές ε, πράξεις. Μετά τη, τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, οι ισχύουσε διατάξει για επιτροπολογία πρέπει να αντικατασταθούν από κατεξιοδότηση πράξη και εκτελεστική πράξη σύμφωνα με δύο άρθρα τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άρθρα 290 και 291. Η προσαρμογή αυτή τη ισχύουσα νομοθεσία τη διατάξη τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχει μεγάλη σημασία, ιδίω για του τομεί εκείνου πολιτική όπω η Αλία, που ρυθμίζονται από διατάξει που δεν υπάγονται στη διαδικασία συναπόφαση, που δεν υπάγονταν μέχρι τώρα στη διαδικασία συναπόφαση και δεν είχαν προσαρμοστεί για τον αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω τη διαδικασία τη ρυθμιστική αρχία με έλεγχο που τέθηκε σε ισχύ μετά το 2006. Εν ώψη αυτών των δύο διαφορετικών διατάσεων, οι συντάκτε ε, ήθελαν να δείξουν σαφέστερα την φύση αυτών των δύο διαφορετικών κατηγοριών πράξεων. Η για τις κατεξιδοτήσεις πράξεις ο νομοθέτης αναφέρει στην Επιτροπή να υιοθετήσει μέτρα μπορεί να αναθέσει ο ίδιος. Άρα ο νομοθέτης πρέπει να ελέγξει αυτή την ε, λειτουργία, την δράση της Κομισιόν. Στα πλαίσια των εκτελεστικών πράξεων, το πλαίσιο είναι διαφορετικό. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης. Οι πράξει αυτέ απαιτούν ενιαίο τόσο τρόπο εκτέλεσης και άρα η Κομισιόν πρέπει να ασχίσει τις εκτελεστικές δραστηριότητε. Άρα τα κράτη-μέλη θα ελέγξουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων, των εκτελεστικών αυτών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Η νέα συνθήκη αναφέρει σαφώ ότι τα κράτη-μέλη και μόνο είναι αρμόδια για τον έλεγχο των αρμοδίτων αυτών της Επιτροπής αν απαιτείται ένας τέτοιος έλεγχος από ένα ε, νομικά δεσμευτικό νομικό κείμενο της, της, της Ένωσης αν και ε, παρότι αυτή η αρμοδιότητα ανήκει στα κρατημέλη, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να έχουν δικαίωμα παρακολούθησης του ενδεδειγμένου τρόπου ε, εφαρμογής της ε, δραστηριότητας αυτής, ιδίως αν η βασική πράξη είναι αρμοδιότητά τους. Οι γνωμοδοτήσεις ΚΟΥΝ έχουν στόχο να θέσουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση στον τομέα των εκτελεστικών πράξεων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον το δικαίωμα που έχει αυτή τη στιγμή ε, για τη διαδικασία επιτροπολογία που συνδέονται με την βασική πράξη που υιοθετείται με βάση τη διαδικασία τη απόφαση. Πρόκειται για το δικαίωμα παρακολούθηση, πρόσβαση εγγράφων κλπ. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου πρέπει να έχουν πρόσβαση στι συνεδριάσει των επιτροπών που περιλαμβάνουν εκπροσώπου των κρατών μελών το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει και τα δύο όργανα να μπορούν να επιφέρουν αντιρρήσει σε ένα σχέδιο εκτελεστικού μέτρου που είναι αντίθετο με την ε, πρόθεση του συνσηγητή. Ένα άλλο σημαντικό θέμα της έκθεσης είναι να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ελέγχει στο μέλλον τις ε, δράσεις επιτροπολογίες που υιοθετήθηκαν πριν τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Το θέμα αυτό ε, είναι σημαντικό, διότι στον τομέα τη αλληλεία δεν υπάρχει άλλη εξουσία στην απόφαση για την έγκριση των νομοθετικών πράξεων. Η Επιτροπή, όπως και οι περισσότερες επιτροπές του Κοινοβουλίου, θεωρούν ότι στο θέμα αυτό, που το ονομάζουμε ευθυγράμμιση, η προσέγγιση δεν πρέπει πρέπει να καλύπτει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα γενικού χαρακτήρα και όχι μόνο τα συγκεκριμένα μέτρα. Είναι εξάρτητα από τον τρόπο λήψη απόφαση, την διαδικασία επιτροπολογία που που εφαρμοζόταν στο μέτρο αυτό πριν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα. Η ευθυγράμμιση πρέπει να γίνεται αναπερίπτωση για να εξασφαλίζει ότι όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα γενική σημασία που εγκρίθηκαν μέχρι τώρα στα πλαίσια των άρθρων 4 και 5 τη απόφαση του Συμβουλίου τη 28 Ιουνίου 1999 που καθορίζουν τι διαδικασίε, του τρόπου εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων που ανακτήφεται στην Επιτροπή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Για να εξασφαλιστεί η εξουσία της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στις εκτελεστικές πράξεις και να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, ο κ. Κούν ζητά από την Κομισιό να θεσπίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα έναν κατάλογο των πράξεων αυτών. Έχω και μια συνθετική, ε, ένα συνθετικό σημείωμα από τον κύριο Κούν. Τι θέλει συνοπτικά το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίζεται ισότιμα από την Κομισιόν ως συνομοθέτης σε όλες τις εκτελεστικές πράξεις και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, το Κοινοβούλιο να διατηρήσει τα, ήδη, τα φυστάμενα δικαιώματα, ιδίω το δικαίωμα παρακολούθησης και εν τέλει το Κοινοβούλιο να μετέχει στις συνεδριάσεις που παρίστανται τα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα τρία βασικά ζητήματα που ζητούμε που ζητά ο κύριο Κούνεξ εξ ονόματός μας. Αυτά. Ε, προφανώς ήταν παθιασμένη η θέση μου και ελπίζω να σας κινητοποίησε και εσάς. Ευχαριστώ, Άλεν. Με βάση τα σχόλια που έκανε στο προηγούμενο κείμενο, με αυτό το κείμενο αποκτούμε νομικά τις αρμοδιότητες να νομοθετούμε. Είναι τεχνικό θέμα. Η Κομισιόν θέλει να σχολιάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Καντέγκ για τη σαφή του παρουσίαση. Δεν θα επανέλθω στη θέση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μία πρόταση όπως είπατε που είναι πολύ σημαντική διότι εφαρμόζει τις νέες διατάξεις της συνθήκης όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις και ο στόχος μας είναι καταρχήν να λάβουμε υπόψη τις καινοτομίες της νέας συνθήκης, ένα νέο δηλαδή θεσμικό πλαίσιο και μέσα στα στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει μια επιτροπολογία πιο αποτελεσματική, πιο απλή, πιο διάφανη από αυτή η οποία ισχύει τώρα. Δεν θα επανέλθω στα θέματα αυτά, απλώς θα ήθελα να τονίσω τα σημεία που τόνισε ο κύριος Καντέκ και που αναφέρονται στο σχέδιο εκθέσεως του κυρίου Κούν. Το πρώτο είναι πώς θα επιλέξουμε μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών επιτροπολογίας. Προτείνουμε δύο, συμβουλευτική και ε, εξετάσεως, όπου ε, θα υπάρχει ενισχυμένος έλεγχος σε σχέση με τη συμβουλευτική. Στην, ε, στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως προτείνεται η, εξέταση να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα γενικά θέματα και να έχει ο νομοθέτης μεγάλη ευελιξία για να επιλέξει την διαδικασία σύμφωνα με ε, τις εκτελεστικές πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πιο αυστηρή θεωρούσαμε ότι η διαδικασία πρέπει να είναι του, του κοινού δικαίου και η ε, μελέτη να περιορίζεται μόνο σε αριθμητικά περιορισμένες περιπτώσεις. Αυτά λοιπόν τώρα θα συζητήσουμε την ε, προσέγγιση της Επιτροπής που θέλει να περιορίσει ε, τον έλεγχο σε ευαίσθητα θέματα αλλά βέβαια υπάρχει υπάρχει ευρία ερμηνεία του ευαίσθητου ε, τομέα οπότε ε, αυτό πρέπει να δούμε. Όσον αφορά την τροπολογία 6β το δικαίωμα της ε, αντιρρήσεως του, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εσείς προτείνετε να αποκαταστήσετε το δικαίωμα εξετάσεως που προβλέπετε τώρα στο άρθρο 8 της Επιτροπολογίας και αντί για απλώς το, Κοινοβούλιο θα συμπεριληφθεί τώρα και το Συμβούλιο για να μπορεί να εφαρμόσει εκτελεστικές πράξεις. Θα ήθελα να σας πω γιατί ε, η Επιτροπή δεν ε, επανέλαβε αυτή τη δυνατότητα εξετάσεως στην ε, πρότασή της. Κατά για να σεβαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο διότι ε, το άρθρο 291 προβλέπει ότι μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να ελέγξουν τις εκτελεστικές πράξεις. Από πλευράς απόψεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να παρέμβει στην εφαρμογή μιας εκτελεστικής πράξεως. Δηλαδή ούτε το Συμβούλιο ούτε το Κοινοβούλιο και γι' αυτό εκεί θεωρούμε ότι είναι ισότιμοι τα δύο θεσμικά όργανα τα οποία δεν μπορούν να μπλοκάρουν μία εκτελεστική πράξη. Μόνο τα κράτη-μέλη έχουν αυτό το δικαίωμα ελέγχου. Γι' αυτό και ένα άρθρο το οποίο θα ονομαζόταν αντίρρηση θα ήταν ουσιαστικά νέο. Αλλά αυτό μήπως σημαίνει ότι δεν έχουν δικαίωμα να σχολιάσουν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι βέβαια, αυτή δεν είναι η δικιά μας ερμηνεία. Εμείς θεωρούμε ότι έχουν δικαίωμα εποπτείας, ε, δικαίωμα ε, μιας ε, εξέτασης το δικαίωμα να επισημάνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να της πούν προσέξτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβαίνετε τις αρμοδιότητές σας, υπερβαίνετε τις προθέσεις του, νομοθέση, του νομοθέτη πράγμα το οποίο είναι ένα δικαίωμα του που υπάρχει αλλά δεν πρέπει να οδηγήσει στο να μπλοκάρει τις διαδικασίες. Δεν μας ενοχλεί ε, η επισήμανση ή η εξέταση αλλά αυτό που είναι αντίθετο στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών είναι το μπλοκάρισμα και το μπλοκάρισμα το οποίο υπάρχει τώρα σύμφωνα με την παλιά συνθήκη έχει ένα μειονέκτημα δηλαδή Τώρα στέλνουμε στο Κοινοβούλιο ε, περίπου 900 εκτελεστικές πράξεις το χρόνο για να εξασκήσει το δικαίωμά του εξετάσεως. Και αυτές ε, οι διαδικασίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν και ε, μας, ε, μας ενημερώνει το κοινοβούλιο μία ή δύο φορές το χρόνο. Δηλαδή ουσιαστικά ε, μπλοκάρουμε διαδικασίες οι οποίες δεν ε, δεν επανεκκινούνται παρά μία ή δύο φορές το χρόνο. Οπότε ε, μπλοκάρουμε και μειώνουμε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι το Κοινοβούλιο να πάση στιγμή έχει δικαίωμα να ενημερώσει την Επιτροπή, να τους πει ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά εγώ δεν συμφωνώ ότι θα έπρεπε ε, να ε, ε, ανακόπτουμε με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή μιας διαδικασίας. Τη μόνη φορά που το Κοινοβούλιο πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ανεκάλεσε μία πράξη ήταν πέρα των δυνατοτήτων ε, εξετάσεως του Κοινοβουλίου. Άρα το Κοινοβούλιο δεν είναι ο μόνος, ε, δεν είναι μόνος αποτελεσματικός τρόπος να βελτιωθεί η διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση. Ίσως οι προσπάθειες δεν είναι επαρκείς και εμείς θα θέλαμε να υποφεληθούμε και να βελτιώσουμε την ε, ενημέρωση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και αποφασίσαμε αποφασίσαμε ε, να ε, καταργήσουμε όλες τις διαφορές μεταξύ συναποφάσεως ή μη. Θα υπάρξει ενημέρωση του Κοινοβουλίου εφεξής για όλα τα θέματα και όλες τις ε, νομοθετικές πράξεις. Τέλος, η ευθυγράμμιση. Ο κύριος Καντέκ μας είπε σαφώς ότι πρέπει να ξαναεξετάσουμε το παρελθόν για να το ευθυγραμμίσουμε με την νέα συνθήκη. Αλλά ακόμη και αν ακριβές αυτό δεν πρέπει να αμφισβητήσει το άρθρο 10 της προτάσεώς μας το οποίο αυτομάτως ε, ε, προβαίνει σε μία ευθυγράμμιση ε, τεχνικά για να αποφύγουμε στο μέλλον να ισχύσει και η παλιά και η νέα επιτροπολογία. Θέλουμε να εφαρμόζεται μόνο η νέα επιτροπολογία σε όλες τις ε, μελλοντικές ε, ε, εκτελεστικές πράξεις. Αυτό το οποίο πολύ σωστά είπατε είναι ότι αν περιοριζόμαστε στο άρθρο 10 θα ξεχνούσαμε τα πεδία τα οποία στο παρελθόν δεν υπησέρχονται εις την συναπόφαση. Πολύ σωστά το Κοινοβούλιο θέτει το θέμα αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να στρεβλώσει το σημείο αυτό την πρότασή του. Σε σχέση λοιπόν με την πρόταση την οποία έχετε στο τραπέζι, εξετάζουμε τώρα την εφαρμογή στη συνθήκη τη Λισαβόνας των νομοθετικών πράξεων που δεν είχαν προηγουμένως ε, ε, εφαρμοστεί όπως η γεωργία, η αλληλεία, ορισμένα θέματα της Γενικής Διευθύνσης ε, ΣΑΝΚΟ γιατί δεν χρειαζόταν εργαζόντουσαν στην Θα ξανεξετάσουμε λοιπόν όλα τα θέματα από πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας για να δούμε αν υπάρχουν τομείς όπου εξουσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα απορρέουν από το άρθρο ο 290 δηλαδή του άρθρου που αναφέρεται στα έργα κατά ανάθεση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπουσέ, πλήρης παρουσίαση της έκθεσης Κουν, όπως είπα, προθεσμία για τις τροπολογίες είναι Παρασκευή, 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία θα γίνει στις 2 Ιουνίου στην Επιτροπή για να παρουσιάσουμε την γνωμοδότησή μας στην Νομική Επιτροπή που θα ψηφίσει 2 και 3 Ιουνίου. Σημείο 7. Εγκρίνουμε τις τοπολογίες στη Σύμβαση για, τις την μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλληλείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού. στόχος είναι να τοποποιηθεί ο κανονισμός 3178 του 78 που υιοθετήθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 78 για την επικύρωση από την Ένωση της Σύμβασης για την ε, πολυμερή, μελλοντική πολυμερή συνεργασία στην στο βορειοτικό Ατλαντικό. Η έκθεση αυτή ανατέθηκε στον κύριο Βαλέντσα από το ΕΛΚΑ στις 7 Απριλίου. Ένας, ε, η πρώτη αυτή παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Την περασμένη φορά δεν είχαμε και πολλούς πολλούς στη συζήτηση. Ούτε τώρα έχουμε πολλούς πολλούς. Προτείνω, επειδή η παρουσίαση δεν είχε γίνει παρόντος του εισηγητή, να ζητήσουμε πρώτα από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να μιλήσει για τα βασικά θέματα της πρότασης και κατόπιν να ζητήσουμε από τον κύριο Βαρένσα να μιλήσει για να κάνει σχόλια. Όπως και τα άλλα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να μιλήσουν η κυρία Κορντέκα της Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σωστά είπατε ότι κάναμε μια προκαταρτική παρουσίαση της έκθεσης αυτής, αλλά με χαρά να σας την ξαναπαρουσιάσουμε. Να σας πω το ιστορικό πλαίσιο του εγγράφου. Όπως ξέρετε, ο, ο Οργανισμός του Βορειοδυτικού Ατλαντικού ε, ιδρύθηκε με μια σύμβαση του 78. που υιοθετήθηκε με, την, ε, με τον κανονισμό του Συμβουλίου που αναφέρεται. Το 78 όμως είναι πολλά χρόνια. Πριν και έκτοτε πολλά πράγματα έγιναν και στην αλληλεία και στον τρόπο διαχείρισης ε, των αλληλευτικών αποθεμάτων. Μην ξεχνάτε επίσης και τη συμφωνία του 1995 για την ε, συμφωνία για τα λαποθέματα, τη συμφωνία του ΦΑΟ, τη συμφωνία για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2002. Έκτοτε τα κράτη-μέλη του ΝΑΦΟ θεώρησαν ότι η σύμβαση δεν ήταν επίκαιρη, δεν εξέταζε, δεν λαμβάνε υπόψη τα νέα εργαλεία και δεν είχε και έπρεπε να τροποποιηθεί. Έκτοτε δημιουργήθηκε ή προχωρήσαμε σε μια σειρά τροποποιήσεων της σύμβασης που λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις αυτές Έχετε λοιπόν αυτό το κείμενο του Συμβουλίου, της αποφάσης του Συμβουλίου που έχετε μπροστά σας. Να σας πω εντάχει τα άρθρα και το τι προσφέρουν στη σύμβαση αυτά τα άρθρα. Οι κύριες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο είναι το άρθρο 1. Περιλαμβάνονται νέοι όροι, αλευτικοί πόροι, αλευτικές δραστηριότητε και περιγράφουν σαφώς τι σημαίνει ο ορισμός αυτός. Δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε ασυνέπειες. Ε, όλοι γνωρίζουμε γιατί μιλάμε, άρα επί από αυτού υπάρχει συμφωνία. Τα άρθρα 2 και 3 περιλαμβάνουν τις νέες αρχές, τις σύγχρονες αρχές διαχείρισης αλίας. Όπως είπα γίνονται, έγιναν πολλές αλλαγές τα τελευταία έτη. Τα άρθρα αυτά αντικατοπτρίζουν λοιπόν τις εξελίξεις. Το άρθρο 5 εξετάζει την απλοποίηση της δομής της οργάνωσης. Τώρα υπάρχουν δύο όργανα λήψη αποφάσεων, το Γενικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Αλληλείας, που δημιουργούν κάποιες δυσκολίες, πρόκειται για μια δομή περιττή πλέον, συγχωνεύτηκαν σε ένα σώμα. Το άρθρο 9 είναι αναθεώρηση του, της φόρμουλας, του τρόπου υπολογισμού της, ε, στον προϋπολογισμό που αντικατοπτρίζει, που αντικατοπτρίζει πλέον το αρχείο και ο χρήστη πληρώνει. Άρα το 60% του προπολογισμού κατανέμεται μεταξύ των συμβαλωμένων μερών ανάλογα με τα αλλιεύματα. Τα άρθρα 11 και 12 περιγράφουν τις ευθύνες του κράτους σημαία και του κράτους λιμένα δίνοντα σαφέστερο τρόπο για τι υποχρεώσει των, ε, από, των αποβιβάσεων. Το άρθρο 13 ε, αλλάζει τον τρόπο λήψη αποφάσεων από πλειοψηφία σε πλειοψηφία 2 τρίτων. Το 14 είναι ένα σημαντικό βήμα μπρο όπου τροποποιούμε τη διαδικασία ε, αντίρρησης. Όταν ένα κράτος ε, διαφωνεί με τη διαδικασία ε, πρέπει να εξηγήσει το λόγο και να πει επίσης τι μέτρα προτίθεται να λάβει συγγνώμη έτσι μπερδεύτηκα από την συζήτηση και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει συμπληρωματικά ως προς το υιοθετηθέν μέτρο. Το 14 δίνει μεγαλύτερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά το άρθρο 15 είναι νέα διαδικασία επίλυσης διαφορών που επιτρέπει ταχύτερη επίλυση των διαφορών. Αυτές είναι οι αλλαγές της σύμβαση εν ολίγης. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Συνάδελφε, πολύ συνοπτικά. Κύριε Βαλέντσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέπετε να παρουσιάσω για δεύτερη φορά το θέμα αυτό. Προς το παρόν έχω μόνο ερωτήσεις και θα υπάρχουν ερωτήσεις κατά τη ε, διάρκεια της την προετοιμασία της Βλέπουμε εδώ ότι η αλλαγή της ε, Convention χρειάζεται πλειοψηφία τριών τετάρτων. Προς το παρόν ποια είναι τα κράτη που έχουν κυρώσει αυτή τη σύμβαση και ποια όχι. Επίσης, γιατί μόνον τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κυρώσει αυτές τις αλλαγές ενώ τα συμβαλόμενα μέρη ήδη το έκαναν το 2007 και το 2008. Επίσης, στο μέλλον, ποια είναι τα, μέσα, τα μέτρα που θα λάβει η Κομισιόν ώστε να μην υπάρχουν ε, στην διαδικασία τέτοιου είδου καθυστερήσει. Επίση, θα κάνω το εξή σχόλιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Αλίας θα πρέπει να εκπροσωπείται στις ε, μελλοντικές ε, διαπραγματεύσεις που γίνονται. Ποτέ δεν είχε ζητηθεί η απόψή μας, η μετοχή μας το 2007 και 2008. Σήμερα όμως βάσει των νέων μας αρμοδιοτήτων κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται. Θα ήθελα να επιθυμίσω στην Κομισιόν ότι είναι υποχρεωμένη να σέβεται τις νέες διαδικασίες και τις νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για κάτι το καινούριο. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Και βεβαίως τα πλαίσια αυτής της διαδικασίας είναι αργά. Αλλά θα ήθελα να πω ότι εφ' εξής θα πρέπει να είμαστε παρόντες σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ τον κύριο Βαλένσο, ο κύριος Γκάλαχερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Η ΝΑΦΟ δεν ήταν, ήταν παρούσα εδώ και πάρα πολλά ε, χρόνια διαπραγματεύσεις όταν ακόμη πολλά σημερινά μέλη δεν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σημερινές ανάγκες και να ληφθεί υπόψη το οικοσύστημα να υπάρχει μεγαλύτερη ευκρίνεια σε αυτά τα οποία λέγονται για τις υποχρεώσεις όλων των μελών και θα ήθελα επίσης να πω ότι για την διαδικασία επίλυσης ε, διαφορών και για οποιαδήποτε άλλη διαξία θα πρέπει να είμαστε παρόντες. Αυτά τα λέω και στα πλαίσια της ε, συνεργασίας, στα πλαίσια της νέας ε, σύμβασης. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν βάσει της κοινή λογική και λαμβάνοντα υπόψη τι ισχύουσε διαδικασία σήμερα. Η Κομισιό, για να απαντήσει σε ερωτήσει του κύριου Βαλέσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξή. Οι χώρες οι οποίες έχουν κυρώσει Υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Μέχρι τώρα όμω πρέπει να πω ότι η Νορβηγία ε, δεν έχει προχωρήσει και η τελευταία χώρα που επικύρωσε ήταν ο Καναδάς από ό,τι μαθαίνω. Πρόκειται λοιπόν για θέματα τα οποία είναι ακόμη εκκρεμή για τις χώρες αυτές, τα πλαίσια της Σύμβασης του Νόφου, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Δανία, καταρχήν στην Γρυλανδία, ασχολείται η Βουλή με αυτά τα θέματα. Γιατί αυτό το θέμα χρόνισε τόσο πολύ στην Κομισιόν. Θα πρέπει να σας πω ότι η γαλλική εκδοχή και οι τροπολογίες της σύμβασης εγκρίθηκαν το 2008. Και μόνο τότε μπόρεσε η Κομισιόν να ασχοληθεί με αυτή την κατάσταση. Επίσης θέλω να σας πω ότι η Κομισιόν είχε κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τα νομικά, σε τη νομική βάση την οποία έπρεπε να καθορίσει. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η πρώτη σύμβαση ενεκρίθηκε με τη μορφή κανονισμού από το Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε απόφαση του Συμβουλίου και βεβαίως τη δεκαετία του 70 τα πράγματα γίνονταν εντός διαφορετικά από ό,τι σήμερα καταλαβαίνετε. Ίσως γι' αυτό ε, έχουν ε, αυτές τις ε, καθυστερήσεις και μετά από ε, διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο βλέπουμε ποια είναι η πιο κατάλληλη διαδικασία σήμερα. Επίσης, όπως ξέρετε, τέθηκε και πρόβλημα με τις γραπτές μεταφράσεις, δεδομένου ότι ο αρχικός κανονισμός ε, κυρώθηκε μόνο στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα. Σήμερα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, θα πρέπει να μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε όμως ότι πρόκειται για μία μακρά διαδικασία. Προφανώς όλες οι γλωσσικές εκδοχές θα είναι από τον Ιούνιο στη διάθεσή μας. Άρα θα έχετε κι εσείς στα πολωνικά αυτές τις τροπολογίες σύμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κι εγώ, λεω Πρόεδρος, για αυτές τις εξηγήσεις. Η παρουσίαση λοιπόν του σχεδίου έκδοσης θα γίνει στις 14 ε, Ιουλίου και η ψηφοφορία στις 30 Αυγούστου. Πράγμα που σημαίνει ότι στην ε, δεύτερη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου θα ψηφιστεί από την ε, Ολομέλεια. Διότι όπως ξέρετε έχουμε δύο περιόδους συνόδου. Λοιπόν, τελειώσαμε με την σημερινή αδάκτηση σήμερα το πρωί. Είχαμε πει το πρωί, όπως ζήτησε η κυρία Ρόντος, ότι θα κάνουμε αν είχαμε χρόνο συζήτηση για το θέμα της πετρελαιοκυλίδας στον κόλπο του Μεξικού. Παρ' όλα αυτά, είχα πει ότι χρειαζόμαστε και κάποιον εμπειρογνώμονα από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να μας εξηγήσει ποιες είναι σε, με μεγαλύτερες λεπτομέρειες οι επιπτώσεις αυτής της πετρελαιοκυλίδας για την αλληλεία και για την ε, εισαγωγή αλληλευτικών προϊόντων. Και η Γενική Διεύθυνση ε, Περιβάλλοντος δεν ε, έχει, είχε χρόνο να το κάνει αυτό. Εάν θέλετε, θα μπορούσαμε το θέμα αυτό να το συμπεριλάβουμε στη μερισσία διάταξη της επόμενης συνάντησης που θα έχουμε και θα ζητήσουμε από την Επιτροπή όντως να μας αποστείλει έναν εμπειρογνώμονα ο οποίος θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις ε, αυτή της μεγάλη προβλήματος, δηλαδή της πετρελοκυρίδας που δημιουργήθηκε στον κόλπο του Μεξικού και των επιπτώσεων που θα έχει για την αλληλεία και για τις εισαγωγές αλληλευτικών προϊόντων. Δεν ξέρω αν θέλει τώρα κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποια πρόταση ή να το αφήσει για την άλλη φορά. Αναφέρεστε στη συνεδρίαση του Στρασβούργου, λέει ο κύριος Γκάλαχερ, ή στην επόμενη συνεδρίαση που θα έχουμε εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ, στις Βρυξέλλες. Γιατί θα πρέπει να, τότε θα έχουμε περισσότερο χρόνο για αυτό το θέμα. Έχει καλώς. Οπότε τελειώσαμε για σήμερα το πρωί και θα